Bonjour à tous. Buenos días. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ενώ είναι τόσο εξαίσιο το πρωινό στις Βρυξέλλες, κάποιοι από τους καλεσμένους μας έχουν δυσκολία να έρθουν στο Κοινοβούλιο λόγω κυκλοφοριακή συμφόρησης. Αλλά πιστεύω ότι ανεξάρτητα από όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε για να εκμεταλλευτούμε τον διαθέσιμο χρόνο με τον επωφελέστερο τρόπο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας σε αυτή την ακρόαση. για το σημαντικό θέμα του ασύλου και της επανεγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο, πακέτο, στο λεγόμενο πακέτο ασύλου Ως πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής ε, Δημοσίων Ελευθεριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλω να σας υπενθυμίσω την σημασία, την μεγάλη σημασία που επέχει αυτό το πακέτο μέσα στην στρατηγική εφαρμογής της ε, συνδίκης της Λισαβόνας και μετατροπής του τρίτου πυλώνα των εσωτερικών θεμάτων σε κοινοτικό, σε ενωσιακό καλύτερα πυλώνα. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρό μετά από το 2009 για να εκφραστεί η πολιτική φιλοδοξία και η συνταγματικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σημαντικό βήμα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την δική μα Επιτροπή, την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Μετά από την θέση εφαρμογή τη ε, Συνδίκη Λισαβόνα, η Επιτροπή μα έχει αναβαθμιστεί και είναι σημαντικός εταίρος στην νομοθετική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, την ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στα κοινά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και φυσικά εμπλέκεται σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση των πολιτών, των ειδικών, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε σαν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ως, ως ε, αλλοδαπή, ως ετούμενοι ασύλου, ως πρόσφυγες, ως άτομα τα οποία επιζητούν προστασία, ως άτομα τα οποία προσπαθούν να διαφύγουν από καταστάσεις απελπισίας. Όλα αυτά έχουν θέσει σε δοκιμασία την ικανότητα της Επιτροπής μας να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα νομοθετικά ζητήματα και σίγουρα τα θέματα τα, τα εσωτερικά, τα θέματα των δημοσίων ελευθεριών, τα άρθρα που καλύπτει από τα άρθρα 67 ως 89 είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία περιλαμβάνουν βασικές ρήτρες όπως η ρήτρα αλληλεγγύης. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση λοιπόν ενώπιόν μας και αποφασίσαμε να την αντιμετωπίσουμε βάσει του σχεδίου το οποίο υιοθετήθηκε μετά τη Σουηδική Προεδρία βάσει του προγράμματο τη Στοκχόλμη το 2009. Πρόκειται για ένα σχέδιο δράση λοιπόν για την υλοποίηση <clears throat> του προγράμματο τη Στοκχόλμη που συνεχίστηκε και από την Ισπανική Προεδρία και τις επόμενες προεδρίες, Ο στόχο είναι μέσα σε πέντε χρόνια να ενσωματωθούν όλα αυτά τα θέματα πλήρω στο νέο σχήμα τη Λισαβόνα. Υπήρξαν <clears throat> μεγάλες δυσκολίες δεν ήταν εύκολο και δεν θα είναι εύκολο και στο μέλλον. Σε ορισμένα από αυτά τα σημαντικά ζητήματα έχουμε καθυστερήσει κάπως σε σχέση με τα σχέδια τα οποία είχαμε κατατήσει καταρχήν. Αλλά έχουμε κάθε υποχρέωση να προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους οι οποίοι έχουν θεσπιστεί μέσα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Και για αυτό το λόγο, με στόχο να επιτείνουμε τον ρυθμό της θεσμικής συνεργασίας για τα θέματα αυτά, έλαβα το λόγο ενώπιον του Ατύπου Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης στην έναρξη της τρέχουσας Πολωνικής Προεδρίας, στην συνεδρία του Σόποτ και θέσα την ιδέα του να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας, διαθεσμικής συνεργασίας μεταξύ της Κομισιόν του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε την ε, υιοθέτηση του πακέτου ασύλου που είναι το πιο προεξάρχον θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα ε, αναγνώρισης ε, και κατάταξης των προσφύγων, Δουβλίνο 2, Eurodac, προστασία, <clears throat> όλα αυτά. Σύνθηκες υποδοχής των, ε, των ετούντων ασύλου και επανεγκατάστασή τους. Όλα αυτά είναι λοιπόν αναπόσπαστα τμήματα του σημαντικού αυτού συνόλου φακέλου, φακέλων και κάθε ένα από αυτά τα θέματα έχει ως αρμόδιο ένα διακεκριμένο εισηγητή στην Επιτροπή μας. Η Πολωνική Προεδρία έχει υιοθετήσει την ιδέα αυτή και έχει δείξει σημαντική προσήλωση για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια μεταξύ Κοινοβουλίου Κομισιών και Συμβουλίου και εμείς από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά της Επιτροπής ε, Δημοσίων Ελευθεριών συμμετέχουμε σε αυτή την ειλικρινή και ανοιχτή συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα ώστε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Και νομίζω ότι έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον ε, Υπουργό τον κύριο ο οποίος εκπροσωπεί την ε, Πολωνική Προεδρία για την προσωπική του δέσμευση και τις προσπάθειές του για να ευδοκιμήσουν αυτές τις προσπάθειες. Είναι πολύ συχνά στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, καταγράφει τις ιδέες οι οποίες διατυπώνται στην Επιτροπή μας και προσπαθεί να τις ενσωματώσει μέσα σε μια γενικότερη συνένεση. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για μια ακόμα φορά για την προσήλωσή του και την ηγετική του δράση μέσα στα πλαίσια των θεμάτων αυτών για να εκμεταλλευτεί και το να τύχει εκμετάλλευση μάλλον το παράθυρο ευκαιρίας μέσα εισαγωγικά που έχει ανοίξει. Μπορούμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε στις συζητήσεις που έχουμε σήμερα αφού σας υπενθυμίσω ότι το υπάρχον κοινοτικό εργαλείο η η δυνατότητα προσωρινής προστασίας δεν έχει ακόμα τύχει τόσο μεγάλης χρήσης μέχρι τώρα και επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της επανεγκατάστασης διότι είναι πιεστικές οι συνθήκες στον περίγυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους έχει προκαλέσει η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη και οι αναταραχές στην ε, νότια οχθή της Μεσογείου Έχουμε λοιπόν ενώπιον μας αυτή την πρόκληση για να δώσουμε σάρκα και ωστά στο άρθρο 80 της Συνδίκης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ρήτρα αλληλεγγύης, ώστε κάθε κάτος μέλος το οποίο είναι υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει διαχείριση κρίσεων λόγω μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσει να βασιστεί και στην αλληλεγγύη των άλλων και να μην αφαιθεί στην τύχη του με όλα τα συμπαροματούντα προβλήματα. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο αριθμό από καλεσμένους ομιλητές και εισηγητές βέβαια για τα επιμέρους θέματα που θα λάβουν το λόγο και να προχωρήσουμε στην ανάλυση των θεμάτων ασύλου και επανεγκατάστασης. και μέσα στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να ευνοήσουμε την επίτευξη συμφωνιών για να ξεπεράσουμε παρεξηγήσεις και δυσκολίες και να εξασφαλίσουμε την ε, καλύτερη ροή πληροφοριών προς όλους τους εμπλεκομένους. Ώστε να αυξηθεί και η αμοιβαία εμπιστοσύνη που είναι και ένας από τους στόχους της Πολωνικής Προεδρίας στο Συμβουλίο των Υπουργών και η οποία έχει αγωνιστεί για να επιτύχει μια πρόθεση των θεμάτων αυτών στο Συμβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον ε, Υπουργό τον κύριο Μίλλερ για την προσωπική του προσήλωση στα θέματα αυτά και του δίνω το λόγο ώστε να ξεκινήσει και η σειρά των ομιλητών όπως προβλέπονται. Κύριε Υπουργέ, Υπουργέ Εσωτερικών Θεμάτων στην Πολωνία. Σας δίνω το λόγο για να παρουσιάσετε την κατάσταση των πραγμάτων όπως τη βλέπει το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω θυμίζοντας ότι τον Ιούλιο του 2011 ο Πρόεδρος ε, υπήρξε ο εισηγητής των τροποποιήσεων του κοινού πακέτου για το άσυλο. Χωρίς ε, την θαραλέα σας πρωτοβουλία, νομίζω ότι θα είμαστε σήμερα σε τελείως διαφορετική θέση όσον αφορά την έκβαση των ε, συνομιλιών μας. Η Πολωνική Προεδρία προσπαθεί να εξεύρει λύση σε, μια, σε ένα δύσκολο συμβιβασμό ανάμεσα στο Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Αυτόν τον συμβιβασμό μπορούμε να τον οικοδομήσουμε με ποικίλου τρόπους, υποβάλλοντας τα μεμονωμένα έγγραφα ε, ε, υποβάλλοντας τα λέω σε διαπραγμάτευση λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις ε, ε, οι διαφωνίες, οι γνώμες που εκφράζονται, ε, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε πολύ γραφειοκρατικές τις συζητήσεις μας. Θα προτιμούσα να γίνεται πραγματική συζήτηση για τα ζητήματα αυτά και για όλα τα προβλήματα που προκύπτουν και που βεβαίως ε, μνημονεύουν ακριβώς την ανάγκη για μιας νέα στρατηγική, ε, ε, μιας νέα εργασίας που θα βασίζεται στο διάλογο. Και κατά αυτήν την έννοια η Πολωνική Προεδρία αποδίδει στο κοινό σύστημα ασύλου πρωταρχικό χαρακτήρα ε, και το καθιστά ένα ζήτημα που είναι προτεραιότητα για τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας ε, και από άποψη ανθρωπιστική, από άποψη ανθρώπινη, αλλά ε, επίσης και ως ανταπόκριση στην ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση που επικρατεί σε διάφορες χώρες μέλη. Γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε, θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε τη δέσμη αυτή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ε, και βεβαίως η μεγάλη πρόκληση παραμένει αυτή η ημερομηνία, η προθεσμία μέχρι το τέλος του 2012 και είναι στίχημα ε, του τρίου της Προεδρίας, της Πολωνικής, της Δανέζικης και της Κυπριακής. Για να επιτευχθεί ο στόχος μας, αυτό τον οποίο ανέφερα προηγουμένως, χρειάζεται μονολυθική συμπαγής πολιτική βούληση. Γιατί διαφορετικά οποιαδήποτε προσπάθεια, οποιαδήποτε δέσμευση, οποιαδήποτε εργασία εμπειρογνωμόνων ή πραγματογνωμόνων από μόνη της δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας και να στέψει με επιτυχία την όλη διαδικασία. Αναφέρθηκα προηγουμένως σε ένα συμβιβασμό. Τούτος ο συμβιβασμός δεν είναι καθόλου εύκολος γιατί ε, ε, υπάρχουν και κάποιες ε, χώρες μέλη, τις οποίες δεν αφορά τόσο πολύ το θέμα του ασύλου. Δεν βαρύνονται δηλαδή τόσο με το βάρος και το κόστος που πέφτει στις πλάτες των χωρών που είναι πρώτες χώρες υποδοχής. Επίσης, δεν επιλέγονται ε, από τους ετούντες άσυλο ε, ισομερός και με ίδιο τρόπο οι χώρες. Ε, δεν είναι χώρες στόχοι των ετούντων άσυλο όλες οι χώρες και εν πάση περιπτώσει γι' αυτό αυτή η κοινή δέσμη μέτρων ε, ίσως για μερικούς δεν είναι απαραίτητο να είναι τόσο κοινή. Μετά από τρεις μήνες κοινή ε, εργασίας και συνεργασίας είχαμε την ε, δυνατότητα να ακούσουμε τους εμπλεκόμενους ε, φορείς. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση των διαπραγματεύσεων, στη στάδιο βρισκόμαστε δηλαδή. Πρέπει να εγκριθεί η οδηγία έτσι ώστε να φτάσουμε ε, σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο όσον αφορά τους πίνακες αντιστοίχησης. Ε, θα ζητηθούν προφανώς ε, και κάποιες διευκρινήσεις από τα θεσμικά όργανα. Πάντω, εμεί ευελπιστούμε ότι οι τροπολογίε, τις οποίες έχουμε, ε, οι τροποποιήσεις μάλλον τις οποίες έχουμε υποβάλει θα γίνουν δεκτές από το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, σε επίπεδο μεμονωμένων ομάδων εργασίας η Προεδρία έχει ήδη προτείνει μια συμβιβαστική λύση η οποία έγινε δεκτή μάλλον ευνοϊκά από τα περισσότερα κράτη-μέλη. Ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ε, επί Πολωνικής Προεδρίας τις συζητήσεις για αυτό ε, ε, το νομικό κείμενο όσον αφορά την Eurodac φέτος το φθινόπωρο υπευλήθη ένα νέο σχέδιο το πιο ακαθόδες ζήτημα είναι η εφαρμογή ε, της ε, συμφωνίας του, ε, του Δουβλίνου βάσει ενός έκτακτου κανονισμού. Στο Συμβούλιο της 22ης Σεπτεμβρίου που συμμετέσχουν όλα τα μέλη, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση αυτού του έκτακτου ε, εργαλείου μέσα στα πλαίσια το, της ε, Συμφωνίας του Δουβλίνου. Πάντως έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερο ε, συζητήσεις για δημιουργία ενός πρώιμου επλοστασίου αντιμετώπισης κρίσεων. Κανένα κράτος μέλος ε, δεν έχει ε, τοποθετηθεί εναντίον αυτής της ε, προτάσεως. Τα κράτη-μέλη απευθύνθηκαν στην Προεδρία ζητώντας αποσαφηνήσεις για τον κάθε μηχανισμό έτσι ώστε να καταλάβουν τον και να προσμετρήσουν την προστιθέμενη αξία της πρότασης. Όσον αφορά τώρα τη διαδικαστική οδηγία, η Προεδρία έλαβε υπόψη της όλες τις συνεδριάσεις των αρμοδίων ομάδων εργασίας που μελέτησαν την οδηγία. Και την 5η Οκτωβρίου η Προεδρία υπέβαλε την πρώτη συμβιβαστική πρόταση. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ε, απομονώσαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα, ε, τα ζητήματα δηλαδή τα οποία θα ε, πρέπει να κοιτάξει η Προεδρία με μεγαλύτερη προσοχή. Επίσης, δεσμευτήκαμε έτσι ώστε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες σε ολόκληρη τη δέσμη, σε ολόκληρο το πακέτο ε, γιατί ας πούμε όταν εσείς κύριε Πρόεδρε προτείνατε οι εργασίες της Επιτροπής ε, Επαφής ε, να συμπεριλαμβάνουν και το Κοινοβούλιο, αυτό είναι μια πολύ σωστή πρόταση. Νομίζω ότι οι τρεις συναντήσεις, συνεδριάσεις οι οποίες έχουν ε, διοργανωθεί εδώ ε, έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα ε, σε αυτήν την προσπάθεια εξέβρεσης λύσης σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Κατά αυτήν την έννοια θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για αυτήν την σημαντική συνδρομή της στην προσπάθεια εξέβρεση συμβιβασμού. και βεβαίως θα συνεχίσουμε την εργασία μας μέχρι τα τέλη του εξαμήνου και ε, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2012 και αν κρατηθεί ο ρυθμός που έχουμε ξεκινήσει, τότε οπωσδήποτε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των τριών αποδοχών, των τριών εγγράφων. Ευχαριστώ. Είναι πολύ καλά τα νέα που μας λέτε. Το γεγονός ότι υπάρχει δέσμευση ώστε να ολοκληρωθεί το θέμα μέχρι το τέλος του 2012 και θα συμμετέχουν και οι τρεις προεδρίες, και η Πολωνική, και η Δανική και η Κυπριακή στη συνέχεια. Είναι πολύ ενθαρρυντική αυτή η προοπτική δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και πολλές ε, επιπλοκές σε όλα τα ζητήματα. Ιδίω εντό του Συμβουλίου. Στη συνέχεια έχουμε την κυρία Μαρία Ασένιους, εκ μέρου της Επιτρόπου Μάλστρομ, είναι προϊσταμένη του Γραφείου της Επιτρόπου, ε, η οποία είναι Επίτροπος υπεύθυνη για θέματα εσωτερικών υποθέσεων. Κυρία Ασένιους, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ να σας διαβιβάσω τους χαιρετισμού της Επιτρόπου Μάλτρομ, η οποία θα ήθελε να βρίσκεται εδώ σήμερα, ε, σε αυτή την τόσο επίκαιρη ε, ακρόαση και θα ήθελα να συγχαρώ και την Επιτροπή σας για τη διοργάνωση. Πλησιάζει το 2012 και αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο ενός κοινού συστήματος ασύλου πριν ε, το τέλος του 2012, τότε δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Η βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ε, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά υπάρχουν ε, εθνικές διαφορές που παρακολύουν την ε, διαδικασία. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Πέρσι πάνω από 50.000 ετούντες άσυλο κατέφτασαν στη Γαλλία, άλλοι τόσοι περίπου και στη Γερμανία και... 35.000 στην Εσθονία. 35 άτομα στην Ιστονία. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μικρά τα ποσοστά. Άλλες χώρες έδωσαν το 44% ενώ η Ιρλανδία έδωσε καθεστώς ε, ε, ασύλου σε 1,6% μόνο. Έχουμε πολλούς ε, ε, μετανάστες από την Τσετσενία και το Ιράκ. Ε, είχαμε ποσοστά αναγνώριση σε κάποιες χώρες μέλη της τάξης του 1, του 2, του 3%, ενώ σε κάποιους άλλους, άλλες χώρες για τους ετήντες άσυλο είχαμε ποσοστά Τη τάξη του 85% ή του 90%. Είναι παράδεκτο να υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές σε, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ε, έχουμε κοινέ αξίες και συμμεριζόμαστε τις ίδιες συμβάσεις, όπως για παράδειγμα τη Σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες που θα ορτάσει τα 60 της χρόνια φέτος. Τι καλύτερο τρόπο λοιπόν από το να γιορτάσουμε αυτή την επέτειο, από το να εγγενιάσουμε μια νέα κοινή πολιτική ασύλου. Οι ανισότητες ε, σήμερα σημαίνουν ότι ε, ουσιαστικά ε, οι ετούντες άσουλο μπαίνουν σε μια κληροτίδα και είναι, ανεξάρτητα από το που καταθέτουν την αίτησή τους τελικώς αποφασίζουν να πάνε σε χώρες όπου θα δεχτούν την αίτησή τους. Υπάρχουν χώρες που δέχονται περίπου το 90% των ε, ε, αιτήσεων. Αυτές είναι οι 10 ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιπες 17 θα πρέπει να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει σαφέστερους κανόνες, κανόνες που θα μπορούν να εφηβερμοστούν από όλους και θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι σημαντικό λοιπόν η νομοθεσία μας να διασφαλίσει ότι οι αιτούντες άσυλο θα τη χάνουν ισότιμης μεταχείρισης οπουδήποτε καταθέσουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν τις ίδιες δυνατότητες διεθνούς προστασίας. Να σας δώσω σύντομα λοιπόν την εικόνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις πιο διεξοδικές προτάσεις, τις συνθήκες υποδοχής. Οι κανόνες ενισχύει αυτή τη στιγμή είναι πολύ ανοιχτοί στην ερμηνεία τους από τα κράτη-μέλη, που σημαίνει ότι οι αιτούντες άσυλο τη σήμερον ημέρα δεν έχουν ε, αντίστοιχη φροντίδα ε, και ε, πρόνοια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και πριν από τρία χρόνια προτείναμε την εναρμόνιση. Ε, ο στόχος είναι να υπάρχει αξιοπρεπής αντιμετώπιση και συνθήκες διαβίωσης για όλους τους αιτούντες άσυλο. Ε, το Συμβούλιο μας είπε ότι είναι πάρα πολύ διεξοδικό το πρόγραμμα και πολύ δαπανηρό και αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος. Ε, η Επιτροπή εισάκουσε το αίτημα και επομένως καταθέσαμε τροποποίηση της πρότασής μας τον Ιούνιο φέτος. Και νομίζω ότι έτσι δόθηκε μια νέα όθηση στις διαπραγματεύσεις και η ακρόαση αυτή το αποδεικνύει. Το άλλο καλό νέο φυσικά είναι η Πολωνική Προεδρία η οποία ε, έχει δεσμευτεί ιδιαίτερα για αυτό το τόσο δύσκολο ζήτημα. Το σκεπτικό μας ε, είναι να ε, αναδιανομηθεί το κόστος για την ε, διαδικασία ασύλου και την οδηγία που κατατέθηκε. Η οδηγία αυτή θέλει να έχει αποτελεσματικούς κανόνες ως προς το κόστος, να αντιμετωπίζονται δυνατότητες ε, για ε, αιτήσει ε, κατάχρησης, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά να είναι ευθογραμμισμένοι με το αναπτυσσόμενο επίπεδο νομολογίας, ώστε να μπορούν να σταθούν και όλα αυτά τα πράγματα στο δικαστήριο. Έχουμε λοιπόν αναδιατύπωση και ταυτόχρονα έχουμε και αναδιατύπωση της οδηγίας για την ποιότητα του ασύλου και αυτή τη στιγμή ήμασταν στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων που είναι πολύ σημαντικό διότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και η ΚΟΡΕΠΕΡ έχουν εγκρίνει τα θέματα αυτά επί της ουσίας και το να τα εγκρίνουμε τελικώς θα δείξει ότι υπάρχει δυνατότητα να συμφωνήσουν τα τρία θεσμικά μας όργανα και φυσικά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε καλύτερα τις διαπραγματεύσεις μας για το υπόλοιπο πακέτο. Έχουμε επίσης τον κανονισμό του Δουβλίνο Όλοι συμφωνούν ότι το σύστημα του Διβλίνου θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού ε, συστήματος ασύλου, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία ως προς το πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Εάν το σύστημα του διβλίνου θέλουμε να είναι εύρωστο, θα πρέπει να ε, θεωρείται από όλους ότι είναι μια δίκαιη λύση και επομένως να το εφαρμόζουν στη συνέχεια. Όσον αφορά το σύστημα του Διβλίνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποστηρίζει την πρόταση της Πολωνικής Προεδρίας ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Θα υπάρχει ένας είδους έλεγχος, ένα health check για να προλαμβάνουμε τα προβλήματα ήδη εκ των προτέρων και αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι δυνατότητές μας και θα υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη για το σύστημα. Θέλουμε να μην υπάρχει ιδιαίτερο άχθος, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να έχουμε ένα καλό σύστημα έγκαιρε προποδοποίηση, αν δεν υπάρχει σοβαρή παρακολούθηση από όλα τα κράτη-μέλη. Σε γενικέ γραμμέ, εξετάζοντας αυτό το πακέτο του ασύλου, νομίζω ότι είναι σαφές ε, σε όλους ότι θέλουμε να αυξήσουμε το συνολικό επίπεδο προστασίας, να ξεφύγουμε από την έννοια των ελάχιστων προτύπων, διότι θέλουμε να αποφύγουμε ε, τον αγώνα προς τα κατώτατα όρια και φυσικά να υπάρχουν κάποιες κοινέ προδιαγραφές. Και υπάρχει και αυτό το οποίο σας ανέφερα νωρίτερα, τα αποτελέσματα που έχουμε από τις ε, ελλείψεις και τις διαφορές που έχουμε από τους τρέχοντες κανόνες είναι πολύ σημαντικά. Ε, σήμερα στη διάρκεια της ημέρας θα συζητήσουμε καθόδη ζητήματα όπως είναι τα θέματα της αποτελεσματικής ε, αντιμετώπισης, τα ε, παιδιά που κάνουν αίτηση ασύλου και όλοι θέλετε να καταλήξετε σε συμφωνία μέχρι το τέλος του 2012. Αλλά Ελπίζω ότι το Συμβούλιο Υπουργών θα μπορέσουν να καταλήξει σε μία απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι στη διάθεσή σας για να σας υποστηρίξει και να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση ε, για όλα αυτά τα ζητήματα, διότι είναι απαραίτητο. Ωστόσο, ένα κοινό σύστημα ασύλου ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών ασύλου και για να έχουμε πρακτικά καλή συνεργασία Υπάρχει πλέον ένα γραφείο υποστήριξης για το άσυλο, το οποίο δρεύει στη Μάλτα. Θα λάβει ε, καθήκοντα πρακτικής καινοτομίας, να υπάρχει η ίδια εκπαίδευση και κατάρτιση ανά την Ευρώπη, ώστε όλα τα γραφεία ασύλου να εργάζονται με τον ίδιο τρόπο. Επίσης θα αξιολογήσουμε πού έχουμε αποτελέσματα, πού δεν έχουμε αποτελέσματα, και φυσικά θα υπάρχουν και εκθέσεις για τη χώρα καταγωγής, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν την ίδια βάση όταν ε, λαμβάνουν αποφάσεις και θα υπάρχουν και ε, δυνατότητες πρακτικής συνδρομής σε χώρες που βρίσκονται υποπίεση. Επίσης θα δημοσιευθεί και μια ανακοίνωση για την ελληνική σύντομα ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ των κρατών μελών που θα περιλαμβάνει τα υφιστάμενα εργαλεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά. Εκ ε, επισημαίνουμε πόσο σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να τηρούν τα ιστορικά τους θέματα σε τάξη. Πριν ζητάτε λοιπόν αλληλεγγύη από τους υπολείπους, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε λάβει και εσείς τα κατάλληλα μέτρα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα πεδίο εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία υποστηρίζεται και από καλές πρακτικές δράσεις, από συνδρομή, από αλληλεγγύη, από παρακολούθηση, αξιολόγηση και ε, δημιουργία δυνατοτήτων και εμπιστοσύνη. Η αλληλεγγύη δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνο μεταξύ των κρατών μελών. Εμεί θα πρέπει να διασφαλίσουμε και αλληλεγγύη και μεταξύ των εταίρων μα και μεταξύ των πιο ευάλωτων ανθρώπων που χρειάζονται προστασία, ιδίω αυτού που βρίσκονται σε στρατόπεδα προσφύγων. Έχουμε και περιφερειακά προγράμματα προστασία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να προχωρήσει περαιτέρω την επανεγκατάσταση ω μία από τι λύσει που προτείνεται για του πρόσφυγες. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το σύστημα επανεγκατάσταση που προτάθηκε ήδη από το 2009 και θεωρώ ότι είναι κρίμα το γεγονό ότι δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για την ελληνική και θα ήθελα να ζητήσω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να βρουν μια λύση επί του ζητήματο μέχρι το τέλο του έτου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να δημιουργήσει περισσότερα κίνητρα για τα κράτη-μέλη για τα θέματα της επανεγκατάστασης μέσω του νέου Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης που θα αντικαταστήσει το ε, υφιστάμενο ταμείο για τους πρόσφυγες από το 2014. Επίσης, ε, ε, να υπάρχουν και ε, συνιστώσεις επανεγκατάστασης σε κάθε περιφερειακό πρόγραμμα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες επί του ζητήματος, αλλά θέλουμε να υπάρχει περισσότερη δυνατότητα επανεγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι προς όφελος και των πιο ευέλωτων προσφύγων, αλλά και των κοινοτήτων που φιλοξενούν προγράμματα περιφερειακής προστασίας και βέβαια μπορεί να ε, μειώσει και τις πιέσεις στα εθνικά συστήματα ασύλου. Τα περιφερειακά προγράμματα είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Μας έδωσαν τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις δυνατότητες των κρατών ε, στα οποία βρίσκονται ε, και οι άνθρωποι βρίσκονται κοντά στις χώρες καταγωγής τους και τις χώρες διέλευσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προγράμματα στην Ανατολική Ευρώπη και θα ξεκινήσουμε και αντίστοιχα προγράμματα στη Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και στην Τινησία ελπίζουμε πριν από το τέλος του έτους και επιπλέον Έχουμε αναπτύξει ένα κέντρο και στο κέρας της Αφρικής που είναι πολύ απαραίτητο για τους ε, ε, πρόσφυγες από την Γένεια και τον Τζιμπουτί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι μέσω των νέων δημοσιονομικών προοπτικών θα υπάρχουν περισσότεροι πόροι για να επεκταθούν αυτά τα περιφερειακά προγράμματα προστασίας και να δημιουργήσουμε και νέα. Εν κατακλείδη λοιπόν κυρίες και κύριοι, έχουμε πολύ ε, δουλειά μπροστά μας ε, για ένα κοινό σύστημα ευρωπαϊκού ασύλου. Πρόκειται για μεγάλη προσδοκία, μεγάλη φιλοδοξία, δύσκολο έργο, αλλά ένα έργο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποια ε, ε, όθηση και από πλευράς Κοινοβουλίου. Και ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να είμαστε περήφανοι για το επιτευγμά μας, μια νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα συνοδεύεται από πρακτική συνεργασία και αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ασένιους, για την επισκόπηση <clears throat> των προσπαθειών που έχουν γίνει από την Κομισιόν και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για να δημιουργήσει τις δυνατότητες για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και φυσικά να βοηθήσει και το Συμβούλιο να ξεπεράσει, να υπερπηδήσει τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί στο σύστημα του Δουβλίνου και στο Eurodac μεταξύ άλλων. Οι επόμενοι ομιλητές τώρα. Και σας υπενθυμίσω ότι το ΙΑΣΟ που έχει αναφερθεί είναι ένα σημαντικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, το, για την παροχή ασύλου. Έχει προσκληθεί στη, συνέλευση αυτή, στη συνεδρίαση αυτή ο εκτελεστικός του διευθυντής, ο κύριος Ρόμπερτ Φίσερ, δεν μπόρεσε να είναι παρόν γιατί κολλείεται και είναι υποχρεωμένος να παραστεί στις ΗΠΑ σήμερα αλλά φυσικά το γραφείο αυτό, η υπηρεσία αυτή έχει προσκληθεί στην ακροασή μας. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Τίνα Ακετόφτ που είναι μέλος της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Πληθυσμού στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και αυτό είναι ένα σώμα το οποίο εμπλέκεται ιδιαίτερα σε θέματα μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν εκ προημίου εάν μας <clears throat> βοηθήσετε να παραμείνουμε μέσα στα χρονικά όρια γιατί στις 10 πρέπει να αρχίσει και το επόμενο τμήμα της ε, συνεδρίασης εσείς και η κυρία Γκάρλικ θα πρέπει να προσπαθήσετε αν μπορείτε να παραμείνετε μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Παρά το γεγονός ότι θα ήθελα και εγώ να χρησιμοποιήσω λίγο χρόνο εξ ονόματος της Συμβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκλησή σας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ευρύτερη συνεργασία στα θέματα αυτά. Πέντε λεφτά δεν θα μου φτάσουν κατά πάσα πιθανότητα. η αύξηση <clears throat> των ετοιμάτων για άσυλο πιέζει κυρίως το νότιο τμήμα της, ε, της ε, Ευρώπης. Ε, θα περίμενε κανείς ότι προέρχονται όλοι αυτοί από την Αφρικανική Ήπειρο, αλλά οι αριθμοί που έχουν παρουσιαστεί στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο τεράστιοι. <clears throat> Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ζητούν άσυλο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πλημμυρίδα το άσυλο είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Όλοι εμπλεκόμεθα, είτε είμαστε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη εξέφρασε πρόσφατα τι ανησυχίε του της για την έλλειψη συνεκτικότητα στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό αποδοχή ποικίλει πάρα πολύ από τη μία χώρα στην άλλη, όπω αναφερθήκε και Το 2010 η Μάλτα, η Λετωνία και οι 100 χώρες είχαν 60, 50 και 44% ποσοστό αποδοχής, ενώ η Ιρλανδία απέριψε 98,4% από το σύνολο των ε, αιτήσεων ενώ η Ελλάδα απέριψε 97%. Υπάρχει λοιπόν τεράστια ποικιλία μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Μαρία Σένιος αναφέρθηκε για το γεγονός ότι είναι σαν να παίζουν σε κάποια λοταρία αυτοί που ζητούν άσυλο. Και είναι γεγονός ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν διαφορετικά την ανάγκη προστασίας αυτών που ζητούν άσυλο. Αλλά ακόμα και όταν βλέπουν τις ίδιες ομάδες ατόμων υπάρχει τεράστια διαφορά. Οι στατιστικές του, της υπάτης αρμοστίας για τους πρόσφυγες δείχνουν ότι η Ισπανία, ότι η Ιταλία δίνει 95% σε αυτού που έρχονται από τη Σομαλία και η Ισπανία μόνο 7%, η Ελλάδα 0%. Αντίστοιχα, 95% των περιπτώσεων έγιναν δεκτέ στην ε, Φιλανδία και 21% μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να καταβληθούν λοιπόν περισσότερε προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Οι προκλήσει όμως είναι να μπορέσουμε να βρούμε ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να υπογραμμίσω και δύο ζητήματα τα οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για την κοινοβουλευτική συνέλευσή μας. Η κατάσταση των γυναικών που ζητούν άσυλο και η κατάσταση των Ρώμα που ζητούν άσυλο. Σε ό,τι αφορά στις γυναίκες, το ψήφισμά του για τα θέματα φύλου σε σχέση με την διαδικασία άσυλου, η Συμβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης τόνισε ότι πρέπει να λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτών των αιτήσεων ασύλου από τι γυναίκε. Οι γυναίκε ζητούν άσυλο για τους ίδιου λόγους, αλλά είναι πολύ συχνότερα θύματα καταδίωξη που οφείλονται στο γεγονό ότι είναι γυναίκες. Ακόμα και αν είναι ο ίδιος λόγος καταδίωξή τους όπως και για του άλλου, μπορεί να ε, εμφανιστεί με διαφορετικό τρόπο όταν πρόκειται για γυναίκες. Η διάσταση του φύλου λοιπόν δεν λαμβάνεται επαρκώς όταν αξιολογεί κανείς τις αιτήσει ασύρου και αυτό θα ήθελα να το κρατήσετε στο μυαλό σας σήμερα που συζητάμε όλα τα θέματα αυτά. Για τους Ρωμά επίσης. Στο ψήφισμά της για τους Ρωμά η Κοινοβουλευτική Συνέλευση τόνισε ότι αν πρόκειται κανείς από ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τύχει ασύλου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωμά οι ομοίοι την χάνουν καταδίωξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάνε στον Καναδά όπου γίνονται αναγνωριστοί ως πρόσφυγες και μπορούν να έχουν προστασία. Ζητά λοιπόν η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης να αναθεωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική ασύλου τη για τα θέματα αυτά. Κάτι ακόμα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ο στόχο τη ισόρροπη κατανομή του φορτίου μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Το σύστημα του Δουβλίνου θέτει ένα υπερβολικό φόρτο στι χώρε που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Στο πρόσθετο ψήφισμά τη, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ζήτησε να υπάρξει κατανομή αρμοδιοτήτων και φόρτου και τόνισε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ότι η αποτελεσματική προστασία των προσφύγων και των ετουμένων ασύλου δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρί να υπάρχει μια καλύτερη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των χωρών όλης της Ευρώπης. Ένα από τα μέτρα για να επιτευχθεί αυτό, αυτός ο στόχος ήταν η έκκληση σε όλες τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης να συμβάλλουν πλήρως στο πρόγραμμα της υπά αρμοστίας του ΟΗΕ για την επανεγκατάσταση των προσφύγων και να δεχτούν επανεγκατάσταση στην Ευρώπη χωρών ε, ε, προσφύγων από χώρες που δεν έχουν ακόμα ε, αντίστοιχη μεταχείριση των προσφύγων. Θα ήθελα τώρα να έρθω στον πυρήνα τη συζήτησής μα. Το να μπορέσουμε να θεσπίσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση θα μα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε σημαντική πρόοδο για την ποιότητα και τη συνεκτικότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται σε σχέση με την παροχή ασύλου, όχι μονάχα <clears throat> στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στα άλλα πρόσθετα 20 κράτη-μέλη του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Το Σύμβουλιο τη Ευρώπη μπορεί και θα πρέπει να συμμετάσχει και να αρρωγεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μια πάγια νομολογία σε σχέση με τα θέματα του ασύλου που δεσμεύουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά την Ευρωπαϊκή Χάρτα και μια σειρά από συστάσει της Υπουργικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Έχει επίσης ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει ότι διακριβώνονται και ελλείψεις πέραν αυτών που διαπιστώνονται από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρακολούθηση λοιπόν από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισμού και υπέρ της ανεκτικότητας και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η σύμβαση επίσης κατά της βίας εναντίον των γυναικών στην, ε, στον οικιακό χώρο είναι και μία βάση για αιτήσει ασύλου, διότι θεσπίζει ένα ισχυρό και ανεξάρτητο μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των κανόνων σε εθνικό επίπεδο. Εγώ υποστηρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτού του μηχανισμούς και να συνεργαστεί με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να εξευρεθούν λύσεις. Το Συμβούλιο της Ευρώπης θα προετοιμάσει επίσης ελάχιστους κανόνες κράτησης για αυτούς που ζητούν άσυλο και για τους ε, μη ε, σε κανονική κατάσταση μετανάστες. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την κράτηση και εναλλακτικέ μορφές κράτηση. Είναι απαραίτητο Είναι απαραίτητο να υπάρξει καλύτερο συντονισμό λοιπόν μεταξύ των διοργάνων για τα θέματα αυτά. Για να κλείσω. Το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου θα έχει επιπτώσεις και πέραν των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καλύψει και τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το να υπάρχει μια, ένα πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό σύστημα είναι προς όφελος όλων μας. Το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου μας δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε πολλά από τα ενδογενή προβλήματα τα οποία συνδέονται με τη διαδικασία ασύλου. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε κυρία Ακετόφτ και προχωρούμε τώρα μετά το Συμβούλιο της Ευρώπης το οποίο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και δεσμεύεται για αυτά τα ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες. Να ακούσουμε τώρα την ε, προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικών και Νομικής Υποστήριξης της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ε, το Γραφείο της Ευρώπης, την κυρία Μάδλιν Γκάρλικ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ ονόματος ε, της ΥΠΑ της Αρμοστίας ε, των ΗΠΑ για τις πρόσφυγες να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι διοργανώνει ακρόαση για το άσυλο. Έρχεται σε πολύ επικαιρή στιγμή, ε, πρόκειται για σημαντική στιγμή για την πρακτική συνεργασία για το άσυλο και έχουμε και σημαντικές συζητήσεις για την αλληλεγγύη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υπουργό Μίλλερ για τον ηγετικό ρόλο που έχει επιδείξει η Πολωνική Προεδρία. Έχουν γίνει εκτεταμένες διαπραγματεύσεις, υπάρχει στο πρόγραμμα ε, περαιτέρω πρόγραμμα για συζητήσεις και συζητώνται όλα αυτά τα σημαντικά θέματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη τη ανανέωση των διαπραγματεύσεων μέσω τη δημιουργία μια ομάδα επαφή ε, ασύλου μεταξύ των θεσμικών οργάνων που θα διευκολύνει τι ε, συζητήσει. Εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό το επίπεδο συνεργασία και προτεραιότητα που δίνεται στα θέματα ασύλου και θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να επιτευχθεί πρόοδο, δεδομένου ότι είναι πολύ περίπλοκα τα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμή, ε, ιδίω για την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και να συγχαρώ ε, και την κυρία Λάμπερτ και όλου του ευρωβουλευτέ που ασχολήθηκαν με το θέμα, καθώ και την Προεδρία. Ε, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ιδίως ε, για τα δικαιώματα που δίνονται σε όσους λαμβάνουν επικουρική προστασία όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου και τη σχετική οδηγία. Ε, χαιρετίζουμε την έκθεση της κυρίας Γκυγιόμ που αποτελεί πολύ σημαντική βάση συζήτησης. Κάποιοι βέβαια εξέφρασαν ανησυχίες για το κατά πόσον η αναδιατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν υιοθετηθεί, θα επιτρέψει να συνεχίσουν κάποια συστήματα ασύλου τα οποία είναι αποτελεσματικά, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα για ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη προστασίας. Επίσης, η αναδιατύπωση τον Ιούνιο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιε από αυτέ τι ανησυχίε και λαμβάνει υπόψη τη και κάποιε σημαντικέ προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσει για την αναδιατύπωση θα δώσουν τη δυνατότητα στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό και να λάβουν υπόψη του σημαντικά από τα κενά που υπάρχει στην οδηγία. Θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει εμεί από πλευρά υπό τη αρμοστία. Το Μάρτιο του 2010 ε, δημοσιεύθηκε μία έρευνα η οποία ανέφερε πολλές σημαντικές ανησυχίες για την πρακτική εφαρμογή της τρέχουσας οδηγίας ε, για τις διαδικασίες ασύλου. Επισημαίνεται το γεγονός ότι χρησιμοποιείται πολλές φορές η ταχεία διαδικασία που σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και ορισμένες φορές δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν καταλήλως οι αιτήσει και δεν υπάρχει και αρκετός χρόνος ε, για τις συνεντεύξεις που χρειάζονται και τα μέτρα που χρειάζονται για τη διεθνή προστασία. Υπάρχουν κάποιες συνεντεύξεις οι οποίες δεν γίνονται με τον ε, αποτελεσματικότερο και πιο δίκαιο τρόπο και ορισμένες φορές οι υπεύθυνοι για τα θέματα ασύλου δεν λαμβάνουν τη δέουσα κατάρτιση και πολλές φορές ε, υπάρχει ε, άρνηση από πλευράς ε, δικαστηρίου και απομακρύνονται οι αιτούντες ίσολο άσυλο πριν από καταφέρουν να καταθέσουν αίτηση έφεσης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικέ πολιτικέ ευαισθησίε για το θέμα αυτό και ελάχιστη πολιτική βούληση για σημαντικέ υψηλέ προδιαγραφέ και υψηλότερε δικρύλες ασφαλείας. Αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικέ αλλαγέ στην οδηγία αυτή, οι οποίε δεν θα οδηγήσουν απαραίτητα σε αύξηση του κόστου ή σε περιττέ αιτήσει ασύλου, αλλά θα αυξήσουν την ασφάλεια ε, και θα επιτρέψουν να έχουμε μέτρα τα οποία θα είναι σωστά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε δυνατότητα ε, για ευέλικτες διαπραγματεύσεις από όλες τις πλευρές. Τώρα, για την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής έχουν ε, ε, εκφραστεί επιφυλάξεις από κράτη-μέλη για το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί το κόστος εάν υιοθετηθεί η προηγούμενη οδηγία. Τώρα η πρόταση που κατατέθηκε τον Ιούνιο έχει εξελιχθεί πολύ σημαντικά και θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο συμβιβασμό. Για την ύπατη αρμοστία υπάρχουν πολύ σημαντικέ πτυχέ τη υφιστάμενη οδηγία, οι οποίε θα πρέπει να τροποποιηθούν το συντομότερο δυνατόν και θα μπορούσε ίσω να βοηθήσει η νέα πρόταση. Το ένα σημείο είναι το θέμα τη κράτηση και χαιρόμαστε που θα συζητηθεί σήμερα το απόγευμα γιατί για την ύπατη αμορμοστία είναι απαράδεκτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη σήμερα ημέρα να υπάρχουν ελάχιστε νομικές διασφαλίσεις για την κράτηση ανθρώπων που μπορεί με να είναι πρόσφυγε και να κρατούνται με τον ίδιο τρόπο οι με ανθρώπου που θεωρούνται ύποπτοι για ε, διάπραξη αδικημάτων και εγκλημάτων και είναι η ζωτική σημασία να υπάρχει νομοθεσία και διασφάλιση και προστασία των ανθρώπων που κάνουν αίτηση ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η Αρμοστία χαιρετίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγγνώμη, που εκφράζεται μέσω της έκθεσης του κυρίου Μασί Πιντάλγκο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε δυνατότητα να τηρήσουμε κάποιες βασικές αρχές στο μέλλον. Παρακολουθήσαμε επίσης και διαπιστώσαμε σημαντικά προβλήματα με το τρέχον σύστημα του Δουβλίνου κάποιες από τις αλλαγές που προτείνονται στην αναδιατύπωση του κανονισμού θα βοηθήσουν κατά την άποψή μας να βελτιωθεί ο κανονισμός. Ε, θα υπάρχουν σαφέστερα κριτήρια και διαδικασίες για τα κράτη-μέλη, αλλά και προς όφελος ε, των ετούντων άσυλο και επίσης ε, θα υπάρχει και δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού αυτού θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε το σύστημα του Δουβλίνου δεν ε, αυξάνει υπερβολικά το άχθος για κανένα κράτος μέλος. Και επίσης το σύστημα θα πρέπει να δίνει πρόσβαση σε όλους όσους κάνουν αίτηση ασύλου για να γίνεται δίκαιη εξέταση των φακέλων τους ε, ε, βάσει και του κανονισμού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν χαιρετίζουμε και τη δέσμευση των συνομοθετών οι οποίοι θέλουν να κάνουν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε συμφωνία για το κοινό σύστημα ασύλου και τα υπόλοιπα μέσα. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για το θέμα αυτό και μπορεί να χρειαστούν και σημαντικοί συμβιβασμοί επί των προτάσεων. Όσον αφορά το σημαντικό θέμα της αλληλεγγύης που ανέφεραν αρκετοί από τους ομιλητές σήμερα, η Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά έχει ε, θέσει υποχρέωση στο κοινοτικό δίκαιο για πολιτικές ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της ευθύνης. Επίσης υποστηρίζουμε και εμείς αυτή τη ε, ε, δέσμευση μέσω προγραμμάτων τα οποία έχουν εφαρμοστεί επιτόπου στα κράτη-μέλη. Στην Ελλάδα, μια χώρα που αντιμετωπίζει πολύ σημαντικέ προκλήσεις σε θέματα ασύλου, η ύπατη αρμοστή θέλει να δώσει ε, και κατάλληλο προσωπικό για αποφάσεις σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο, να αναπτύξουν ε, ε, υλικό για στοιχεία για τη χώρα καταγωγής και χαιρετίζουμε και την δέσμευση του Γραφείου Υποστήριξης για το Άσυλο και Παρακινούμε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να δίνουν βοήθεια στην Ελλάδα ώστε να μπορεί να δράσει με αποτελεσματικό τρόπο. Η υπαταρμοστία έχει υποστηρίξει και προγράμματα επανεγκατάσταση από τη Μάλτα, μια χώρα που επίση πιέστηκε ιδιαίτερα από του πρόσφυγε και τα τελευταία χρόνια έχουμε και πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την ποιότητα του ασύλου και σε χώρες οι οποίες ε, έχουν σχετικά νέα αλλά και σε χώρες που έχουν σχετικά ε, σταθερά συστήματα ασύλου. Ε, θέλω να υλοποιήσουμε επίσης και ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 12 χώρες ε, για την ποιότητα του ασύλου ε, έγιναν εργασίες για τη βελτίωση και την αύξηση των δυνατοτήτων ε, των γραφείων ασύλου ε, και τη δημιουργία βιώσιμων μηχανισμούς ποιότητας ασύλου στα γραφεία αυτά και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ε, πρωτοβουλίες αυτές, τις οποίες χαιρέτησαν ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη, παρουσίασαν πολύ σημαντικά ε, στοιχεία για τη βελτίωση των θεμάτων ποιότητας και εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να ε, κάνουμε προσπάθειες για τη βελτίωση στα κράτη-μέλη. Και ακούσαμε ότι αυτό θα το αναλάβει και το Γραφείο Υποστήριξης ε, στο μέλλον. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που οι πρωτοβουλίες ποιότητας έχουν συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό και στο ε, πρόγραμμα εργασίας του γραφείου για το 2012 και ελπίζουμε να υπάρξει και κατάλληλη χρηματοδότηση ώστε το θέμα της ποιότητας να αποτελεί βασική προτεραιότητα και στα κράτη-μέλη αλλά και στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον. Θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης ότι είναι πολύ σημαντική η πρόκληση της αλληλεγγύης με τρίτες χώρες. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς, αλλά είναι και μια επονίδιστη αλήθεια. Το γεγονός ότι η, ε, ε, τα ε, οι καταβλισμοί προσφύγων βρίσκονται σε χώρες που δεν έχουν τον εξοπλισμό για να εξυπηρετήσουν πρόσφυγες και σε κάποιες περιοχές του κόσμου που πολλές φορές ε, είναι ήδη χώρες οι οποίες βρίσκονται σε ένοπλη σύραξη ή σε πολύ άσχημες συνθήκες. τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λαμβάνουν συλλογικά πολύ λιγότερους πρόσφυγες από αυτές τις τρίτες χώρες. Επομένως, η αλληλεγγύη με αυτές τις χώρες δεν είναι μόνο ηθική προσχώρη υποχρέωση για όσους υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα εθνικής προστασίας, αλλά είναι και μία από τις βασικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επισημαίνουν πόσο σημαντική είναι αυτή η εξωτερική διάσταση σε πολιτικές ασύλου και μετανάστασης. Υπάρχει ανάγκη για πιο συγκεκριμένη και συνολική αλληλεγγύη σε χώρες που χρειάζονται χρειάζονται διεθνή προστασία και αυτό προέκυψε σαφέστερα στην ε, περίπτωση των ε, προσφύγων από τη Σομαλία. Σε πολλά κράτη-μέλη οι Σομαλοί πρόσφυγες αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των ετούντων άσυλων, αλλά είναι ελάχιστοι σε σχέση με αυτούς που υποδέχονται οι όμορες χώρες της Σομαλίας. 184.000 Σομαλοί έφτασαν στην Αιθιοπία, στην Κένια και στο Τζιμπουτί. Από αυτούς οι 46.000 έφτασαν τις πρώτες τρεις εβδομάδες του Ιουλίου η ΥΠΑ και άλλοι επισήμαναν πόσο σημαντικό είναι ανάγκη να υπάρξει διεθνής υποστήριξη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ε, και την έκκληση αυτή ε, εισάκουσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποια κράτη-μέλη. Όμως ε, επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη υπό τη μορφή δυνατοτήτων επανεγκατάστασης. Υπάρχουν ε, αρκετοί πρόσφυγες οι οποίοι είναι ευάλωτοι και εκτίθενται σε διωγμούς ε, ή σε σοβαρές απειλές και είναι τόσο μεγάλες αυτές οι απειλές που μόνο μέσω επανεγκατάστασης μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή και βιώσιμη λύση. Ε, μέχρι του δε η, ε, τα όσα έγιναν για το θέμα της επανακατάστασης των Σομαλών ήταν ελάχιστα. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία επίσης με τρίτες χώρες και στα θέματα Βορείου Αφρικής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι ευαισθησίες προέκυψαν φέτος όταν αρκετά ε, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να φεύγουν από τις χώρες της Βορειοαφρικής ε, για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι οι αλλαγές οι οποίες οδήγησαν σε αυτή τη μετακίνηση των πληθυσμών μπορεί να βοηθήσουν να έχουμε μακροπρόθεσμα βελτιώσεις στις χώρες αυτές. Και η ευημερία και η σταθερότητα στις χώρες αυτές θα πρέπει ε, να αποτελεί στόχο. Δύο από αυτές τις χώρες, η Αίγυπτο και η Τινησία, είχαν πολύ μεγάλες αφήξεις από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια των σειράξεων ε, υποδέχθηκαν περίπου ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους. Πολλοί από αυτούς έφυγαν σε άλλες χώρες, αλλά κάποιοι από αυτούς παρέμειναν και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονταν βοήθεια και ε, χώρο στέγασης. Πάνω από 5.000 εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στα σύνορα της Λιβύης ε, στα, με την Τινησία και ε, μέχρι ε, τις 30 Σεπτεμβρίου 2.600 πρόσφυγες ε, είχαν δοθεί σε χώρες επανεκατάστασης. Ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα. Η επανεκατάσταση αυτών των ανθρώπων που είναι μικρή στον αριθμό τους ε, θα ελπίζουμε να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να διευκολύνουμε την ανάπτυξη της δυνατότητας προστασίας στην περιοχή. Η επανεγκατάσταση στα κράτη μέλη σαφώς θα πρέπει να ενισχυθεί και από σαφέστερες και πολιτικές ε, ε, οι οποίε είναι υπέρ της υποστήριξης και θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την, την επανεγκατάσταση μέσω του προγράμματος επανεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία χαιρετίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ε, συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα επ' αυτού και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να υπάρχει ένας κατάλληλος συμβιβασμός στο εγγύς μέλλον που θα βοηθήσει να ε, υπερκεράσουμε τις θεσμικές μας διαφορές και να έχουμε ένα νέο μέσο προστασίας το οποίο θα μπορούσε να σώσει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων στο μέλλον. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργάνωσε τη σημερινή ακρόαση και προσβλέπω σε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το πάνελ για τις παρατηρήσεις, τις εισηγήσεις και τις παρατηρήσεις που ε, μας ε, έκαναν. Ε, βέβαια, όσοι ήθιστε εδώ στην Επιτροπή μας, έχουμε λίγο αργοπορήσει. Έχουμε πάντα ημερήσεις διατάξεις που είναι πάρα πολύ ε, γεμάτες ε, και συνήθως ε, αργοπορούμε, είμαστε λίγο πίσω. Εν πάση περιπτώσει βλέπω ήδη τον κύριο Μπουζουτήλ που έχει σηκώσει το χέρι του. Παρακαλώ οι προτάσεις, οι ερωτήσεις συγγνώμη να είναι σύντομες έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να πούμε. Ε, έχουμε μια σειρά πολύ σοβαρών ε, πάνελ. Σε λίγο μάλιστα θα πάρει τη θέση μου η κυρία Τζιν Λάμπερτ ε, και θα προεδρεύσει του επόμενου πάνελ, μετά η κυρία Σεσίλια Βίκστρομ, μετά η κυρία Σιλβί Γκυγιόμ. Το απόγευμα η κυρία Μόνικα Λουίζα Μακοβέη, ο κύριος Αντώνιο Μασίπ και ο κύριος Ρούι Ταβάρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για μια σειρά από κύκλους συζητήσεων ε, που θα ασχοληθούν με επιμέρους ζητήματα του ασύλου και της μετεγκατάστασης. Και επομένως ε, Ελπίζω ότι η κάθε ερώτηση θα αφορά το συγκεκριμένο πάνελ που μόλις έχουμε ακούσει. Κύριε Μπουζουτήλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σε ε, όλους όσους ε, μίλησαν ε, πριν από λίγο στο πάνελ. Νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες και όχι μόνο, πολύ περισσότερο, βλέπουμε ότι χωρίς ε, μηχανισμό αλληλεγγύης δεν θα επιτύχουμε καμία ε, νίκη όσον αφορά αυτή, αυτό το πακέτο ε, για το άσυλο. Εδώ και χρόνια είναι ένα θέμα που ταλανίζει την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τον Δεκέμβριο του 2008, πριν από τρία ολόκληρα χρόνια, είχε προτείνει την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Το Κοινοβούλιο έδωσε άμεσο σήμα λέγοντας ότι στηρίζει την τροποποίηση υλοποίηση του πακέτου. Δυστυχώς όμως το Συμβούλιο δεν κινήθηκε περαιτέρω. Είναι γεγονός επίσης ότι η Επιτροπή πολύ αργά τελικά εκπώνησε αυτήν την ε, ανακοίνωση που έβγαλε φέτος. Νομίζω ότι εάν είχε κινηθεί γρηγορότερα θα είχε βελτιωθεί η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι θετικό που βλέπουμε ότι η Πολωνική Προεδρία πραγματικά θέλει να αρπάξει τον τάβρο από τα κέρατα και θέλει να ε, προσπαθήσει να βρει λύση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε ακόμα να είμαστε ε, αισιόδοξοι γιατί πρέπει να δείξουμε ελληνική για μια σειρά λόγων τους οποίους κατέδειξαν και οι ομιλητές. Ε, αλλά το άρθρο 70 είναι σαφές. Αναφέρει ρητά ότι η κοινή πολιτική ασύλου θα πρέπει να βασίζεται σε μοιρασμένη ευθύνη ε, και σε αλληλεγγύη. Και θα μπορούσα να σας δώσω και άλλους λόγους. Να κάνω όμω κάποιε συγκεκριμένε παρατηρήσει, οι οποίε πιστεύω ότι είναι σημαντικέ όσον αφορά το θέμα τη αλληλεγγύη. Πρώτον, εάν ε, πρέπει να ενταχθεί στην ε, οδηγία του Δουβλίνου ή όχι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό έτσι με θρησκευτική ευλάβεια. Το ζήτημα είναι να λυθούν τα προβλήματα εντός ε, Δουβλίνου, εκτός Λονδίνου, ε, Δουβλίνου με χωριστό <laughs> εργαλείο ε, γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι είναι γενός άδικο ε, το να ε, μεταφέρουμε μονάχα στο, στους ώμους των κρατών που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το βάρος ανθρώπων που τελικά θέλουν μόνο να περάσουν από εκεί και να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μηχανισμός αλληλεγγύης θα είναι υποχρεωτικός ή εθελοντικός συζητήσεις επί συζητήσεων. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα δεσμευτικό μηχανισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν με νοιάζει και τόσο εάν τελικά θα είναι υποχρεωτικός ή εθελοντικός, αρκεί να λειτουργεί. Και ε, μέχρι σήμερα ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ε, για την Μάλτα, τη χώρα μου, πιλωτικό πρόγραμμα σε θελοντική βάση, το οποίο δυστυχώς δεν λειτουργήσε και λυπάμαι που το λέω. Ε, κατέληξε στην ε, μετεγκατάσταση 300 ανθρώπων ε, στις 15.000 που έφτασαν στην Μάλτα. Και βεβαίως αν δούμε το ποσοστό των μετεγκαταστάσεων που πέτυχε η Αμερική, που δεν έχει καμία υποχρεωτική ας πούμε ε, νομοθεσία γι' αυτό, τότε πραγματικά θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει ε, να συζητηθούν όλα τα θέματα αυτά με όλες τις χώρες και περισσότερο και με τις χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, ε, θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και με τις τρίτες χώρες. Αναφέρθηκε το θέμα αυτό. Η Τουνησία δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία από την οποία πέρασε, αυτή την επανάσταση, τις τεράστιες αλλαγές ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να μοιραστούμε τις ε, ευθύνες ε, και με τις χώρες αυτές. Χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν από την Λιβύη. Εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι στριμώχνονται στα σύνορα Λιβύης στην Ισία και η Ευρώπη δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Ο κύριος Μασίπ, σύντομα κύριε Μασίπ αν μπορείτε. Ναι κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να αναφερθώ και στο, στην εκπρόσωπο της κυρίας Μάλστρομ και στην Πολωνική Προεδρία που έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία στα θέματα αυτά. Ήμουν χθε σε μια συνεδρίαση με την Πολωνική Προεδρία για να αντιμετωπίσει τα θέματα που ανέφερε και η Πάτη, η Πάτη Αρμοστία. Και έχω μια έκθεση για τα θέματα αυτά ο ίδιος. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατάσταση που είναι πάρα πολύ θετική, αυτή την θετική όθηση της Πολωνικής προεδρία για να μπορέσουμε να κλείσουμε το ταχύτερο δυνατό αυτό το θέμα και να μην το αφήσουμε να τρενάρει μέχρι το 2012. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία να πείσουμε και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου τα οποία διστάζουν. Και αυτό τονίστηκε και από την Πολωνική Προεδρία και από την πάτη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το πακέτο ώστε να υπάρξει μια πρόθεση στα θέματα αυτά και θέλω να ευχαριστήσω και την Πολωνία για τη θετική της αντιμετώπιση στα ζητήματα αυτά. Θα πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε το πρώτο πάνελ της κυρίας ε, Λάμπερτ, αλλά αν θέλετε να απαντήσετε κύριε Μίλλερ στα σχόλια αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προς την Πολωνική Προεδρία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στα σχόλια του κυρίου Μπουσουτήλ, γιατί νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα εύστοχα. Δεν πρόκειται για τυπικές διαδικασίες το αν θα πρέπει να ενσωματωθεί δηλαδή η αλληλεγγύη στο μηχανισμό του Δουβλίνου ή κάπου αλλού. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, αυτό το οποίο έχει πραγματική σημασία μέσα στα πλαίσια αυτής της συζήτησης είναι το να ληφθεί υπόψη η, η ιδέα αλλά και η ουσία της αλληλεγγύης γιατί αυτό ελείπει αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω ότι ζούμε σε δύσκολες εποχές από πλευράς προϋπολογισμών. Υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα πέραν της αλληλεγγύης που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως ότι ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι θέμα μονάχα χρημάτων. Αν απολέσουμε από τους οφθαλμούς μας την αρχή της αλληλεγγύης, θα χάσουμε την έννοια της αλληλεγγύης για πολλά χρόνια. Θα φύγει και θα ξαναγυρίσει. Συμφωνώ μαζί σας λοιπόν. Ας εξασφαλίσουμε ότι αυτή η θεμελιώδης αρχή γίνεται σεβαστή, η αρχή της αλληλεγγύης. Πάρτε το παράδειγμα της Μάλτας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε <clears throat> έχουν εδώ το πάνω χέρι. Μας έδειξαν ότι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και ότι η ευαισθησία είναι πολύ σημαντικότερη από τις τυπικές διαδικασίες. Εγώ υποστηρίζω το να συζητήσουμε τα θέματα της αλληλεγγύης, αλλά αυτό πρέπει να είναι αποτέλεσμα εσωτερικών συμφωνιών μεταξύ από μεταξύ προσεγγίσεων που έχουν εγωιστικό χαρακτήρα και προσεγγίσεων που θέλουν μια γενική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Λοιπόν, έχει κλείσει επομένως το πρώτο τμήμα της ακροασής μας, που ήταν οι εναρκτήρες παρατηρήσεις. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο πρώτο πάνελ του οποίου θα προεδρεύσει η κυρία Τζιν Λάμπερτ, η εισηγήτριά μας. Σας ευχαριστώ όλους. Σας παρακαλώ να μείνετε όλοι στην αίθουσα για να συνεχίσουμε το έργο μας. Ευχαριστώ. Thank you. We'll be in touch.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 Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το δεύτερο πάνελ. γιατί ήδη βρισκόμαστε, ε, έχουμε αργοπορήσει και επομένως ε, για τους τέσσερις ομιλητές ε, θα χρειαστούμε σαφώς πάνω από 20 λεπτά. Λοιπόν, λέγομαι Jean Lambert και είμαι εισηγήτρια από την πλευρά του Κοινοβουλίου όσον αφορά ε, την ε, οδηγία για τα επαγγελματικά ε, προσόντα. Και, αλλά δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα. Βλέπουμε εδώ στο πάνελ ότι το θέμα είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, ειδικά δε θα γίνει αναφορά στα ευάλωτα άτομα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ε, να δούμε εάν τα ευάλωτα άτομα παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες, πώς μπορούμε να ταυτοποιήσουμε ε, τα ευάλωτα άτομα, ε, τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν έτσι, ειδικές ανάγκες ή ιδιαίτερες ευαισθησίες. Θα πρέπει να τους εφερθούμε με τον τρόπο που φερόμαστε στο γενικότερο πληθυσμό ή με κάποιον πιο ειδικό τρόπο. Έχουμε ήδη ακούσει ότι όσον αφορά τα ευάλωτα άτομα είναι πολύ ευάλωτα και όσον αφορά τη μετεγκατάσταση κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αυτά διεξοδικά. Έχω την τιμή να προεδρεύω ενός εξαιρετικού ε, πάνελ και είναι και πολύ καλό κιόλας που θα ακούσουμε στο Κοινοβούλιο νέες φωνές. Αυτό είναι εξαιρετικό. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Φιλίπ Ντεμπρουχέρ, ε, ο οποίος ε, είναι συντονιστής ακαδημαϊκού δικτύου Έχουμε την κυρία Βαλεντίνο Ντάτ, συντονίστρια για θέματα ισότητα φίλων του Γραφείου του Γενικού Επιτρόπου για του πρόσφυγε και του απάτεδε στο Βέλγιο, τον κύριο Σέλβαν, που είναι δικηγόρο, εμπειρογνώμων για τα δικαιώματα ε, ασύλου ε, για τους ε, LGBTI, δηλαδή λεσβείες, ομοφιλόφιλους, αμφιφιλόφιλους και τρανσεξουαλικά άτομα καθώς επίσης και τον κύριο Ζερόμ Μπογιάτ, ο οποίος είναι διευθυντή ανάπτυξη της οργάνωσης Parkour Dexil, μέλος του Διεθνού Συμβουλίου Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίου, γιατί και αυτό ε, είναι ένα πάρα πολύ ειδικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να μελετήσουμε και να δούμε οπωσδήποτε στα πλαίσια του πακέτου για το άσυλο. Ε, κύριε Ντεμπρούχερ, παρακαλώ, θα είστε ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση λαμβάνοντας ε, υπόψη και την ε, καθυστέρηση που έχουμε όσον αφορά το πρόγραμμα, θα είμαι σχηματικός και πάρα πολύ λακωνικός, ε, γιατί προτιμώ άλλωστε να εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να περνάει καλύτερα το μήνυμα. Λοιπόν, πρέπει να σας μιλήσω για τα ευάλωτα άτομα, τα άτομα τα οποία έχουν ειδικέ ανάγκες που βεβαίως αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι πολύ συχνά ε, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τις ε, καταχρήσεις ε, της διαδικασίας ασύλου, αλλά ξεχνούμε ότι υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχουν ειδικέ ανάγκες, ανάγκες τις οποίες όμως δεν καταφέρνουμε ε, να ε, αντιμετωπίσουμε μέχρι τώρα. Και όσο πιο ειδικέ είναι οι ανάγκε των ατόμων αυτών, όσο πιο ευάλωτα είναι τα άτομα αυτά, τόσο πιο άμεση θα πρέπει να είναι η δική μα ανταπόκριση. Πέντε πολύ σύντομα στοιχεία, ή ε, σημεία μάλλον πρώτη ε, γενιά οδηγιών. Στην ουσία ε, είχαμε μία διάταξη ε, στην, στην οδηγία για την υποδοχή, το άρθρο 17, που έμεινε όμως κενό γράμμα δυστυχώς. Δεν εφαρμόστηκε, διότι πολύ συχνά ερμηνεύτηκε από τα κράτη-μέλη με κάποια κακή πολιτική ε, βούληση. Ε, ε, ξέρετε ότι εάν κανείς αρχίσει να ερμηνεύει τα, τον νόμο, τότε τα πράγματα δεν είναι πολύ θετικά. Όσον αφορά την δεύτερη γενιά, της προτάσεις της Κομισιόν για τις νέες οδηγίες και η πρώτη και η δεύτερη ανασύσταση που αφορά τις συνθήκες υποδοχής και όσον αφορά και την διαδικασία διαδικασία εμείς εξετάσαμε ε, στην, ε, στο ακαδημαϊκό δίκτυο, ε, εξετάσαμε λέω αυτές τις προτάσεις και έχουμε γενικά να δώσουμε ένα θετικό πρόσημο σε αυτές τις προτάσεις του Ιουνίου 2011. Ξέρω ότι συνήθως όλοι κρίνουμε και κατακρίνουμε ε, τις αναπλάσεις των οδηγιών λέγοντας ότι όπως δρομούν είναι ένα βήμα προς τα πίσω. Εμείς όμως αυτή τη φορά θα κάνουμε εξαίρεση και θα πούμε ότι πραγματικά είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τα εμπρός. Τρία σημεία επί της ουσίας τώρα. Πρώτον, ο ορισμός, δέλημα του, του οριζόντιου χαρακτήρα της οδηγίας και της συνοχής επομένως της οδηγίας. Τρίτον, το πρόβλημα της ταυτοποίησης των ενδιαφερομένων. Πρώτον, ο ορισμός. Μιλάμε για ευάλωτα άτομα τα οποία έχουν ειδικέ ε, ανάγκες ή εξειδικευμένες ε, ανάγκες. Συχνά συμβαίνει, έχει ήδη συμβεί δηλαδή επανειλημμένα, τα διάφορα θεσμικά όργανα τα οποία αφορά το κείμενο αυτό ε, να μπερδεύουν τις έννοιες δεν ξέρουμε λοιπόν αν μιλάμε για ευάλωτα άτομα, αν μιλάμε για άτομα ε, που έχουν ειδικέ ανάγκες, ε, αν είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες ή μία. Ε, εάν δεν ορίσουμε σαφώς περί ποιων ατόμων μιλούμε, εάν δεν είναι λοιπόν ο ορισμός τεχνικός και πλήρης, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Νομίζω ότι τώρα έχουμε προοδεύσει θεωρώντας ότι το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο ευάλωτος χαρακτήρας του ατόμου και υπάρχει σχέση αιτίου του ανάμεσα στο ευάλωτο άτομο και τις ειδικέ ανάγκες που έχει. Βεβαίως δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Ε, υπάρχουν ακόμα εδώ και εκεί διάφορα προβλήματα αντίληψης, ας πούμε, ε, οι διατάξεις ε, στην δεύτερη ανάπληση όσον αφορά τις διαδικασίες δεν είναι πάρα πολύ σαφείς. Επίσης, θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα όταν σε κάποιες ε, ε, διατάξεις προβλέπεται αυτοματισμός, δηλαδή ορίζουμε κάποια άτομα ως ευάλωτα και συμπεραίνουμε, τεκμέρουμε ότι παρουσιάζουν και ειδικέ ανάγκες. Αλλά ας πούμε όλα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, όλοι οι ηλικιωμένοι δεν έχουν απαραίτητα ειδικέ ανάγκες. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν τεκμέρονται ε, ε, ε καταστάσεις γιατί μπορεί ε, οι επιπτώσεις όσον αφορά το κόστος βεβαίως να είναι σημαντικές. Ε, δεύτερο σημείο, όσον αφορά τον ηρωζόντιο χαρακτήρα των ε, κειμένων, δηλαδή αυτά τα διάφορα κείμενα τα οποία συζητούν τα θεσμικά όργανα έχουν υπάρξει πρόοδοι. Όμως, ακόμα παραμένουν κάποια προβλήματα. Υφίστανται λοιπόν ακόμα προβλήματα. Στην αρχική οδηγία, η οποία ε, συμφωνήθηκε σε πολιτικό επίπεδο, η διάταξη η οποία εγκρίθηκε, το άρθρο 20 δηλαδή, στην ουσία αναπαράγει το λάθος του άρθρου 17 της πρώτης οδηγίας όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής και μπορούμε να φανταστούμε ότι ε, οπωσδήποτε ε, θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτήν τη νέα οδηγία και θα πρέπει και υποψιαζόμαστε ότι ενδεχομένως θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίστηκε το άρθρο 17. Δεύτερο στοιχείο. Μας προβληματίζει που δεν ε, χρησιμοποιούμε την έννοια του ευάλωτου ατόμου ε, στο, στα πλαίσια του Δουβλίνου. Δεν γίνεται δηλαδή, δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά ε, σε άτομα ευάλωτα, σε άτομα τα οποία παρουσιάζουν ειδικέ ανάγκες και επομένως αυτό μας ενοχλεί γιατί θα έπρεπε να υπάρχει μια, ένας οριζόντιος χαρακτήρας. Τρίτον, η ταυτοποίηση Πρόκειται για ένα ουσιώδες, θεμελιώδες θέμα. Δεν θέλουμε απλώς να καθορίσουμε τα ευάλωτα άτομα. Θα πρέπει και μεταξύ των ετούντων άσυλο να ταυτοποιηθούν ε, τα άτομα αυτά τα οποία παρουσιάζουν ειδικέ ανάγκες. Αυτό προϋποθέτει μια ειδική διαδικασία ή έναν ειδικό μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να ε, υλοποιηθεί έτσι ώστε να ε, γίνεται άμεση αξιολόγηση της κατάστασης των ειδικών αναγκών, του κόστους, της παρακολούθησης κτλ εάν θέλουμε να δώσουμε περαιτέρω εγγυήσει στα ευάλωτα άτομα, οπωσδήποτε θα πρέπει να υλοποιηθεί μηχανισμός ταυτοποίησης αυτών των ατόμων. Βεβαίως έχουν υπάρξει πολλές ε, πρόοδοι γιατί, στην, ε, γιατί πλέον στο κείμενο αναφέρεται ρητά αυτό το οποίο υπενοείται στο άρθρο 17 ε, και επομένως ε, κατά αυτήν την έννοια μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία. Επίσης ε, στη διαδικαστική οδηγία υπάρχουν θετικά στοιχεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι συνάδελφοί μου θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για τα θέματα αυτά αλλά ας πούμε ένα, ένας που ζητάει άσυλο και ο οποίος έχει υποστεί βασανιστήρια ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να εκφέρει έναν λογικό λόγο, έναν ορθό λόγο. Επομένως θα πρέπει ε, να πούμε ότι πραγματικά υπάρχουν πρόοδοι, αλλά όμως η διατύπωση θα πρέπει να χτενιστεί ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισημία. Επίσης, η προβληματική της ταυτοποίησης σε βάθος χρόνου, σε διάρκεια χρόνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ταυτοποίηση του ευάλωτου ατόμου είναι ε, κάτι ευαίσθητο, κάτι δύσκολο και δεν είναι μία ταυτοποίηση η οποία μπορεί να γίνει άμεσα, δηλαδή από την πρώτη ακρόαση του ετούντος ε, άσυλο. Ε, δεν έχει προβλεφθεί κάτι πάνω σε αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί έτσι ώστε να δοθεί ευκαιρία ταυτοποίησης για τους ανθρώπους αυτούς για τους οποίους το ευάλωτο της κατάστασής τους θα εμφανιστεί λίγο αργότερα μετά την πρώτη ακρόαση. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω κυρία Πρόεδρε, μονάχα ε, ένα τελευταίο επί του οποίου θα ήθελα να επιμείνω, είναι γενικού χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό δίκαιο ε, του ασύλου εισάγουμε την ιδέα ε, του ευάλωτου ατόμου. Είναι μια νομική ιδέα η οποία δεν έχει μελετηθεί παρά μόνο ας πούμε στο κοινωνικό δίκαιο και ε, σε, ε, στο φορολογικό δίκαιο ε, για, το άσυλο είναι η πρώτη φορά που, γίνεται, που εισάγεται αυτή η έννοια. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταβάλουν μια προσπάθεια και μια διανοητική αν θέλετε διαδικασία έτσι ώστε να κατανοήσουν πλήρως τι σημαίνει αυτή η έννοια του ευάλωτου ατόμου. Ε, ε, έχουν γίνει προσπάθειες αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν πιο ε, συγκεκριμένες και διαρθρωμένες προσπάθειες έτσι ώστε η αντίληψη να είναι σαφής η οποία θα οδηγήσει σε, μια ένα συγκεκριμένο μηχανισμό ταυτοποίησης που βεβαίως με τη σειρά του σημαίνει ότι θα υπάρξουν, θα προκύψει κάποιο κόστος και καταλαβαίνω ότι λαμβάνοντας υπόψη και την παρούσα οικονομική κρίση οπωσδήποτε πρόκειται ε, για ένα σημαντικό ζήτημα. Ε, εδώ σας ε, παρουσίασα στην ουσία τον ε, καρπό των εργασιών που έκανα μαζί με μία βοηθό η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ ε, σήμερα μαζί μας ε, και με χρηματοδότηση και από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και βάσει της μελέτης αυτής εκπονήθηκε ένα βιβλίο το οποίο θα δημοσιευθεί μέχρι το τέλος του 11 στις εκδόσεις Λαρσιέ. Αυτό ήταν το διαφημιστικό μου σποτ λέει ο μιλητής. Ε, αναμένοντας όμως αυτό το βιβλίο, ε, σας υπενθυμίσω ότι ε, έχουμε κάνει ήδη μία μελέτη για την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ το τέλος του 2010 και ήδη εκεί αφιερώνουμε σημαντικό αριθμό σελίδων σε αυτήν την έννοια των ευάλωτων ατόμων, των ατόμων με ειδικέ ανάγκες και βεβαίως στο βιβλίο που σας δείχνω τώρα ε, δεν είναι ενημερωμένο το υλικό αλλά εάν καμιά βραδιά δεν μπορείτε να κοιμηθείτε αντί να μετράτε προβατάκια Πάρτε αυτό το βιβλίο των 500 σελίδων και ενδεχομένως θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε. Ελπίζω να ήμουν αρκετά σύντομος και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεμπρουκέρα. Και ξέρετε λοιπόν ποιο βιβλίο θα βάλετε στη λίστα για τα δώρα των Χριστουγέννων τώρα. Πάντως ε, το έγγραφο το οποίο σας έδειξε στο τέλος ο κύριος ε, Ντεμπρουχέρ είναι δωρεάν ε, διαθέσιμο έξω από την αίθουσα. Ε, βεβαίως το θέμα της συνοχής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πολύ στο Κοινοβούλιο. Ε, οριζόντιος χαρακτήρας των διατάξεων συνοχή μεταξύ των προβλεπομένων κτλ. Να καλωσορίσω τώρα την δεύτερη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Βαλεντίνα Οντάτ η οποία εξειδικεύεται σε θέματα ισότητας φύλων, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Επιτρόπου για τους πρόσφυγες και τους απάτριδες του Βελγίου. Βλέπετε ότι το ρολόι αμήλικτα προχωράει, οι δείκτες προχωρούν αμήλικτα. Ε, σας δίνω το λόγο λοιπόν, αλλά έχετε λίγο το νου και στο ρολόι. Ε, καλημέρα κυρίες και κύριοι θα ήθελα να εστιάσω την παρουσίασή μου στην ομάδα των γυναικών, ε, κυρίως δε στις ε, ε, γυναίκες οι οποίες ετούνται άσυλο βάσει ακριβώς του φίλου τους. Δουλεύω, όπως γνωρίζετε πλέον, στο γραφείο του Γενικού Επιτρόπου για τους πρόσφυγες του Βελγίου ε, και είμαι υπεύθυνη για θέματα ε, ασύλου βάσει ε, θεμάτων ισότητας φύλων ή λόγω θεμάτων ισότητας φύλου. Πολύ σύντομα θα σας εξηγήσω ποια, ποιο είναι τι κάνουμε εμείς στα πλαίσια του Γραφείου του Γενικού Επιτρόπου για τους Πρόσφυγες. Θα σας δώσω λοιπόν δύο συγκεκριμένα παραδείγματα για να απεικονίσω ειδικέ ανάγκες και ειδικέ περιπτώσεις. Και μετά ε, θα σας πω πώς εμείς στο Γραφείο του Γενικού Επιτρόπου αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία συνδέονται ε, με το φύλλο. Ε, γιατί είναι ένας πολύ εύγλωτος τρόπος για να δείξουμε με ποιο τρόπο ανταποκρινόμαστε εμείς σε αυτές τις ανάγκες τις οποίες έχουμε σε μια πρώτη φάση ταυτοποίηση το Γραφείο Γενικού Επιτρόπου Προσφύγων και Απατρίδων απάτριδων, συγγνώμη, ε, το ΣΕΖΕΡΑ δηλαδή, ε, έχει έδρα το Βέλγιο, έχει δημιουργηθεί εδώ στο Βέλγιο και στα πλαίσια αυτού του γραφείου υπάρχει συντονισμός για θέματα ισότητας φύλων. Είναι ε, αυτό που εμείς ονομάζουμε το κύτταρο για, το, για την ισότητα των φύλων. Είμαστε 12 που δουλεύουμε για το κύτταρο αυτό, προσπαθώντας να εναρμονίσουμε τις πρακτικές και βεβαίως να βελτιώσουμε τις πρακτικές έτσι ώστε το σύνολο των συναδέλφων που αποτελούν το γραφείο του Γενικού Επιτρόπου, 300 περίπου υπάλληλοι, να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προβλήματα σχετίζονται με την ισότητα των φύλων. Πρώτα λοιπόν προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε ε, τους, ε, ε, τους ενδιαφερόμενους. Στα πλαίσια της εργασίας μας στο ΣΕΖΕΡΑ ερχόμαστε ε, σε τακτική επαφή με διάφορα σωματεία ε, βελγικά και ε, δουλεύουμε πολύ και με ένα σωματείο το οποίο λέγεται SOS Νέοι, SOS Jeune. Ασχολούνται κυρίως δε στην και το SOS Βιόλ ε, που, είναι, που αφορά νέους η πρώτη περίπτωση και βιασμούς ε, η δεύτερη περίπτωση δεν έχει να κάνει ε, με τους ετούντες άσυλο αλλά βλέπουμε ότι ο φόβος της επανάληψης αυτής της τραυματικής εμπειρίας, της τραυματικής επίθεσης είναι ίδιος Και ε, πραγματικά ε, είναι ζητήματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ. Ε, πρόκειται λοιπόν για ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερα ευά... βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και επομένως εμείς πρέπει να καταβάλουμε ειδική προσπάθεια έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τα άτομα αυτά, να προετοιμάσουμε και την αποθεραπεία τους κατά κάποιο τρόπο. il se fait qu'il y a un nœud, une difficulté telle que ε, πολύ συχνά οι, τα άτομα αυτά βλέπουμε ότι δεν καταφέρνουν καν να απομονώσουν το πρόβλημά τους, να μιλήσουν γι' αυτό, ε, να εκφραστούν για την κατάσταση την οποία ε, αντιμετωπίζουν. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει ε, τυπολογία ε, την οποία θα μπορούν να ακολουθήσουν ε, όσοι ασχολούνται με τους, ετούντος, τους ετούντες άσυλο έτσι ώστε να μπορέσουν να απομονώσουν από μόνοι τους αν θέλετε τα ευάλωτα άτομα, μια και εκείνα δεν είναι σε θέση να εκφράσουν το πρόβλημά τους. Πολύ σύντομα τώρα θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω την τυπολογία στην οποία έχουμε καταλήξει στο ε, ΣΕΖΕΡ ε, ε, με ενδεικτικό χαρακτήρα βεβαίως έτσι ώστε συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με τους φακέλους των ατόμων αυτών να ξέρουν γιατί πράγμα μιλάμε, να ξέρουμε εάν τα άτομα τα οποία, των οποίων το φάκελο έχουν μπροστά τους έχουν υποστεί ε, κάποιο, ε, κάποια δίωξη ή κάποια βία. Ε, θα, εμείς λοιπόν έχουμε μία τυπολογία η οποία αφορά όλες τις διώξεις που οφείλονται στον γενετήσιο προσανατολισμό στον οποίο θα αναφερθεί ο κύριος Έλβαν μετά, τα εγκλήματα τιμής, τους ακροτηριασμούς γενετικών οργάνων, υποχρεωτικούς γάμους κτλ. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιος ετών έχει αυτό το προφίλ, τότε ε, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Εδώ θα ήθελα τώρα να φτάσω στο δεύτερο σημείο μου, ε, το οποίο αντικατοπτρίζει λίγο αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στο πρώτο πάνελ. Ε, θα πάρω το συγκεκριμένο παράδειγμα των ακροτηριασμών γεννητικών οργάνων γυναικών. Εμείς δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο ε, μοιράσαμε σε 12 χώρες σε σχετικά ε, με την πρακτική των κρατών όσον αφορά το προφίλ των θυμάτων ε, ακροτηριασμών γεννητικών οργάνων. Φτάνουν λοιπόν εδώ γυναίκες μαζί με τις κόρες τους ας πούμε γιατί φοβούνται ότι οι κόρες θα υποστούν κλειτοριδεκτομία αν μείνουν στις χώρες τους σε πολλές χώρες σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, ε, άμεσα ε, η αίτηση θα, ε, θα, θα μπει υπό το καθεστώς της συνθήκης της Γενέβης. Άλλες χώρες λένε εξαρτάται, θα δούμε την περίπτωση, ενδεχομένως θα δώσουμε την δευτερεύουσα βοήθεια. Ε, θα δουλέψουμε και με την συνθήκη της Γενέβης αλλά και με άλλες ε, πρακτικές. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα χωρών, ε, η οποία μάλλον θα, δεν θα δώσει καθεστώς πρόσφυγα, αλλά δευτερεύουσες προστασίες. Μία άλλη ομάδα χωρών λέει ότι ενδεχομένως θα δώσει αυτό το ε, καθεστώς δευτερεύουσας ε, βοήθειας ή ένα ακόμα πιο εξειδικευμένο ε, καθεστώς, όχι όμως το καθεστώς του πρόσφυγα βάσει της συνθήκης της Γενέβης δεν ξέρουν, ε, υπάρχουν και χώρες οι οποίες δεν ξέρουν και ακριβώς γιατί ο κριτηρισμός των, ε, των ε, γενετικών οργάνων των γυναικών αποτελεί πραγματικά έτσι μια βίαιη πρακτική και κάνει τα άτομα αυτά ιδιαίτερα ευάλωτα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια ετούσα άσυλο σε αυτή την κατάσταση είναι εξαιρετικά διαφορετικός από χώρα σε χώρα. Τώρα φτάνω στο πρακτικό σκέλος ε, είπα προηγουμένως ότι θέλουμε ε, να, θέλαμε να βρούμε μία μεθοδολογία ε, έτσι ώστε από τη μία πλευρά να ταυτοποιήσουμε τις περιπτώσεις, από την άλλη πλευρά να δώσουμε λύσεις ή πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ε, και πρέπει να σας πω ότι έχω φέρει μαζί μου τα σχετικά έγγραφα τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ε, ε, άκρη της αίθουσας. Πάντως, αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορούν να επιλέξουν οι αιτούσες άσυλο αν θέλουν η ακρόασή τους να γίνει από άνδρα ή γυναίκα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών επιλέγουν γυναίκα για την ακρόαση. Επίσης θα πρέπει να είναι μόνες τους, έστω και αν στην αρχή λέει ότι ε, δεν υφίσταται οποιαδήποτε δίωξη, ε, παρόλα αυτά και αν συνοδεύεται και το σύζυγό της, παρόλα αυτά θα πρέπει η ακρόασή της να γίνει χωρίς την παρουσία του συζύγου ή χωρίς των άλλων συνοδών. Ε, επίσης ε, θα υπάρχει και η δυνατότητα βρεφονιπιακού σταθμού, ενδεχομένως αυτό είναι ανεκδοτικού χαρακτήρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες αυτές την ώρα της ακρόσης να ξέρουν ότι τα παιδιά τους είναι κάπου ε, ασφαλή κτλ. Επίσης, ε, ήδη το γεγονό ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ε, ομάδα, αυτό το κύτταρο δράση για θέματα τη ισότητα των φύλων ήδη ε, είναι σημαντικό και βεβαίως διαρκώς δουλεύουμε πάνω στα θέματα αυτά. Τώρα είναι τελευταίο σημείο, δεν έχουμε πολύ χρόνο βεβαίως, αλλά να σας πω ότι σας έχω φέρει εδώ ε, ε, ένα εγχειρίδιο το οποίο δημοσιεύσαμε πρόσφατα ε, σχετικά έχει κυκλοφορήσει σε εννέα γλώσσες, θα το βρείτε και αυτό έξω από την αίθουσα. Εκεί αναφέρουμε διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάσουν οι γυναίκες ή τα νεαρά κορίτσια τα οποία ζητούν άσυλο, τις παραπέμπουμε επίσης σε όλες τις οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Ε, οργανώνουμε πολύ, σε πολύ τακτικά διαστήματα επαφές, συνεργασίες με τις οργανώσεις αυτές, ανταλλάσσουμε πληροφορίες έτσι ώστε να, να είμαστε πάντα ενημερωμένοι και έτσι ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς την τυπολογία μας. Ευχαριστώ, πολύ. πολύ. Όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα θέματα των διαδικασιών βλέπουν ότι είναι σημαντικά αυτά τα οποία αναφέρετε. Η κυρία Γκυγιόμ είναι αυτή που θα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και επίσης είναι σημαντικό αυτό που λέτε για την πολυγλωσία στην πληροφόρηση. Ενδιαφέρον ιδίω σε μια χώρα όπως το Βέλιο. Περνάμε στον κύριο Τσέλβαν, ο επόμενος που είναι ο επόμενος ομιλητής μας, είναι δικηγόρος και ο οποίος ασχολείται με τα θέματα των λεσβιών, των ομοφιλοφίλων, αμφιφίλων κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση να λάβω το λόγο ενώπιον του Κοινοβουλίου για τα θέματα των λεσβιών, των ομοφιλοφίλων, των αμφιφίλων, των ε, τρανσεξουαλικών ατόμων και τα θέματα που έχουν να κάνουν με το άσυλο στην Ευρώπη. Το 2007 στη Ζιοζακάρτα υπήρξε μια συνδιάσκεψη της διεθνής κοινότητας συγκεκριμένα για τα θέματα αυτά που άπτονται της ε, ταυτότητος, της σεξουαλικής ταυτότητος και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτό αφορά το, τη δυνατότητα του κάθε ανθρώπου να βρει μια συγκινησιακή και συναισθηματική σχέση με άτομα άλλου ή του ίδιου φίλου παραπάνω από ενός φίλων. Επομένως, δεν βλέπουμε μοναχά θέματα συμπεριφοράς, βλέπουμε και θέματα ταυτότητας για όλα αυτά τα άτομα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα με τον υπολογιστή. Mm. Θα συνεχίσω μέχρι ότου διορθωθεί αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Για την ε, ταυτότητα του φίλου, εμείς θεωρούμε ότι αυτή είναι αυτό το οποίο νιώθει το κάθε άτομο σε βαθύτερο επίπεδο, ποια είναι η δική του εμπειρία του φίλου, που μπορεί να μην αντιστοιχεί με το φίλο το οποίο του έχει αντιστοιχηθεί στη γέννησή του ή με τα χαρακτηριστικά του σώματός του. Μπορεί το άτομο αυτό να έχει ζητήσει ή να έχει επιτύχει τροποποίηση των χαρακτηριστικών, των σωματικών του χαρακτηριστικών για να φέρει σε αντιστοιχεία αυτό το οποίο αισθάνεται με το σώμα του. Εντάξει. Βλέπουμε λοιπόν θέματα τροποποίησης της σωματικής εμφάνισης ή της σωματικής λειτουργίας για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα. Επομένως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν μας ενδιαφέρουν μονάχα οι χειρουργικές διαδικασίες. Το φύλλο μπορεί να μην, το ε, φαινοτυπικό φύλλο μπορεί να μην αντιστοιχεί στη σεξουαλική ταυτότητα. Δεν θέλουμε λοιπόν να εστιάσουμε σε ένα σύνολο ερωτήσεων το οποίο θα αντιμετωπίσει επιτυχώς τις αιτήσει αυτών των ατόμων. Θέλουμε να έχουμε ένα διαφορετικό μοντέλο. Εγώ βλέπω την ταυτοποίηση της διαφοράς για τους ε, ζητώντας ετούντες ασύλο από αυτή την κοινότητα και εδώ αντιμετωπίζουμε και το θέμα του στιγματισμού που προέρχεται από τη σχέση με την οικογένεια, με το κράτος κτλ. Το αίσθημα ε, ντροπή που νιώθουν τα άτομα αυτά και την ε, ζημία που υφίστανται αυτά τα άτομα από την καταπίεση αυτή. Το 2010 το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έδωσε σε μια σημαντική απόφαση κατεύθυνση για τους ζητούντες ασύλου από αυτήν την κοινότητα. Είναι η περίπτωση του Λόρδου Ρότζερ που αφορά τα άτομα τα οποία βρίσκονται στην κατάσταση αυτή και που ουσιαστικά ξεπερνάει αυτή την αντιμετώπιση ότι είναι διαφορετική η συμπεριφορά των λεσβιών και ομοφιλοφίλων από αυτών των ανθρώπων που είναι ετεροφιλόφιλοι. Η βασική όμως ιδέα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα όλοι να ζουν ελεύθερα χωρίς φόβο και να μην υφίστανται καμία ζημία λόγω της σεξουαλικής τους προτίμησης. Όπως το ίδιο ισχύει και για την προστασία λόγω θρησκείας ή φιλετικής προέλευσης. Θα πρέπει όλοι να έχουν τη δυνατότητα να ζουν ελεύθερα χωρίς φόβο καταδίωξης. Αυτό δίνει λοιπόν και κάποιες κατευθυντήρες γραμμές και στην Ευρώπη, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί μας ενδιαφέρει η δυνατότητα να ζει κανείς ελεύθερα χωρίς να υφίσταται διώξεις ή παρενοχλήσεις. Το Σεπτέμβριο του 1900 2005 υπήρξε και μία ε, διακήρυξη που έγινε στο Άμστερνταμ για τα άτομα αυτά που είναι ε, λεσβείες, ομοφιλόφιλοι κτλ. Ξέρουμε ότι είναι πολλοί τέτοιοι ετούντες άσυλοι που ζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Οι συστάσεις του σχεδίου κατά της ε, ομοφιλοφοβίας είναι να υπάρξει και η κατάργηση των νόμων που απαγορεύουν την επαφή ατόμων με το ίδιο φύλλο. Ξέρουμε ότι και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν περάσει ένα ψήφισμα το οποίο αφορά αυτή την αντιμετώπιση και ξέρουμε ότι και στην Αυστραλία φέτος η συνέλευση των κρατών της πρώην κοινοπολιτείας θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά. Ο στόχος μας να εξασφαλίσουμε να υπάρχει αυτή η προστασία και να μην υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ποινικοποιούν τη συμπεριφορά των ατόμων αυτών. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει μια διαδικασία ε, απόκρυψης και δεν θα πρέπει τα άτομα αυτά να καταφεύγουν σε ψέματα και σε σιωπή για να επιβιώσουν. Αυτό ήταν μια σιωπή 10 δευτερολέπτων. Για τα άτομα στα οποία αναφέρομαι δεν αναφέρομαι ούτε σε 10 δευτερόλεπτα, ούτε σε μια εβδομάδα, ούτε σε ένα μήνα, αλλά για όλη τη ζωή. Όλη τη ζωή ζουν σε καθεστώς σιωπή. Και αυτό είναι σημαντικό όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αντιμετωπίσει την περίπτωση Y, που είναι μια προδικαστική αίτηση από την Γερμανία σε περίπτωση προσιλητισμού, θα πρέπει να αναφέρει ότι κανένα άτομο δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι θα πρέπει να απόσχει από δραστηριότητε που βρίσκονται στην καρδιά της ταυτότητάς του. Το σχέδιο αυτό λέει ότι η αυτοταυτοποίηση θα πρέπει να είναι επαρκής για να θεσπίσει την ταυτότητά του. Για τα τροτά λοιπόν άτομα θα πρέπει να είναι αρκετό αυτό. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για την προέλευση των ατόμων αυτών. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τις λεσβίες γιατί αντιμετωπίζουν τεράστια κοινωνική πίεση και κατακραυγή. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα προστασία στα κέντρα υποδοχής. Από την πλευρά του Ευρωπαίου νομοθέτη, νομίζω ότι θα πρέπει να συγχαρούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρξουν και προσφυγές βάσει σεξουαλικής ταυτότητας στο άρθρο 10. Τι περαιτέρω όμως πρέπει να γίνει. Εμείς κατανοούμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν πιο θετικά πρότυπα βάσει του άρθρου 10 όταν λέει ότι η σεξουαλική, σεξουαλικός προσανατολισμός μπορεί να θεωρηθεί λόγος προστασίας μιας ομάδας. Εμείς θα πρέπει να πούμε θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους λόγους προστασίας και η σεξουαλική ταυτότητα. Θέματα ανησυχίες όπως θέματα, για θέματα παιδοφιλίας θα πρέπει να βασιστούν ότι διεθνώ δεν αναγνωρίζεται η παιδοφιλία ως μια έγκυρη μορφή σεξουαλικού προσανατολισμού. Και τα παιδιά τα οποία ε, αναγνωρίζονται ως λεσβίες, ε, ομοφιλόφιλοι κτλ. δεν τη προστασία αυτή τη στιγμή λόγω των νόμων σε σχέση με την ηλικία συνένεσης. Τα παιδιά θα πρέπει να ταυτοποιούνται ως μέλη αυτής της κατηγορίας γιατί είναι ιδιαίτερα τότε. Δεν είναι θέμα σεξουαλικής πράξης, είναι θέμα ταυτότητας. Θα πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνεται λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας ένα άτομο σε μια, στον κατάλογο των ανθρώπων που είναι τρωτά. Ας δούμε τα εξής όμως σημεία. Στις διαδικασίες συνέντευξης για την ταυτοποίηση των ατόμων αυτών υπάρχουν πραγματικά προβλήματα σε σχέση με την ε, αποκάλυψη των ε, στοιχείων τους και την ανάγκη να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα, ασφαλές, σε ένα ασφαλή χώρο. Η περαιτέρω ε, η, εμπειρία που έχουμε συλλέξει δείχνει το πόσο μεγάλη είναι η τραυματική εμπειρία αυτών των ατόμων. Τα άτομα αυτά έχουν αναγκαστεί όλη τη ζωή να κρύβουν ποιοι είναι. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό γιατί είναι πολλά τα κράτη-μέλη τα οποία εμποδίζουν τις αιτήσει των ατόμων που είναι ομοφιλόφιλες, βίες κτλ. Γιατί θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχαν υποβάλει αίτηση επιβάλλει επί τη βάση άλλων ε, στοιχείων. Είναι γεγονός ότι τα άτομα αναγνωρίζουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα μόνο όταν νιώθουν ασφαλείς. Είχα ένα πελάτη ο οποίος ήταν μεταφιλικό άτομο που ήρθε από το Πακιστάν και βιολογικά θεωρείται γυναίκα γιατί έχει αλλάξει φύλο. Αυτό όμως αντιμετωπίζει, οδηγεί σε τεράστια προβλήματα βίας που υφίσταται στα κέντρα κράτησης και από την πλευρά του φίλου του και από την πλευρά της σεξουαλικής ταυτότητας. Οικογένειες. Ο ορισμός της οικογένειας βάσει του Δουβλίνο 2, η οδηγία για την υποδοχή και η οδηγία για την αναγνώριση θα πρέπει να συμπεριλάβουν την πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην περίπτωση Σάφενκοφ που διευρύνει την έννοια της οικογενειακής ζωής για να περιλάβει και ζευγάρια ιδίου φύλου. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει δεχθεί τους ορισμούς και τις αποφάσεις του, του Δικαστηρίου του Στρασβούργου σε σχέση με θέματα που έχουν να κάνουν με οικογένειες και σε ζευγάρια ιδίου φύλου. Όλα αυτά πρέπει να εφαρμόσετε λοιπόν μέσα στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Για να κλείσω λοιπόν, θα πρέπει να διορθώσουμε μια, ένα ιστορικό σφάλμα. Η σύμβαση για τους πρόσφυγες ήταν απόρρια των φρικοδών γεγονότων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα στατόπεδα συγκεντρώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν όχι μοναχα Εβραίοι, αλλά και ομοφιλόφιλοι άνδρες οι οποίοι εξοντώθηκαν λόγω της σεξουαλικής ταυτότητας. Το 1981 έφερε, ήρθε το θέμα αυτό στα Ολλανδικά δικαστήρια, 1991 στα Αγγλικά δικαστήρια. Είναι καιρός αυτή η προστασία όμως να δοθεί όχι μοναχα μεμονωμένα, αλλά σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σαφήνεια των ε, λόγων σας. Και είναι ενδιαφέρον για όλους τους ε, ομιλητές μας να δίνουν συγκεκριμένες αναφορές στα θέματα στα οποία αναφέρονται. Προχωρούμε τώρα στον Ζερόμ Μποαγιάτ που είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστήριων και τίθεται και πάλι το θέμα της αναγνώρισης των ειδικών αναγκών που αναφέρθηκε προηγουμένως Ζερόμ. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν αυτά τα οποία μας πεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο σήμερα. Είμαι διεθνή ανάπτυξη της Parcours d'Exil που είναι μέλο του Διεθνού Συμβουλίου Αποκαταστημάτων Βασανιστήριων. Είναι ένα φορέα στο Παρίσι που αντιμετωπίζει τα θύματα βασανιστήριων. Έχουμε περίπου 650 άτομα τα οποία είναι υποπερίθαλψη στο κέντρο μας. Είμαστε μέλος του Διεθνού Συμβουλίου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστήριων, που είναι ένας ανεξάρτητος φορέας χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το 1 τρίτο των κέντρων για την αποκατάσταση βασανιστήριων είναι στην Ευρώπη και είναι κυρίω φορεί τη κοινωνία των πολιτών που δρούν για την πρόληψη των βασανιστήριων και την αποκατάσταση των θυμάτων. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα θύματα έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα κέντρα αποκατάστασης, έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να συμβάλλουμε στην πρόληψη των βασανιστήριων. Περίπου 100.000 με θύματα βασανιστήριων αντιμετωπίζονται κάθε χρόνο από τους φορείς αυτούς. Ο οργανισμός αυτός, το Διεθνές Συμβούλιο Αποκατάστασης, έχει πολυπίκυλα μέλη. Υπάρχουν κέντρα που αντιμετωπίσουν χιλιάδες θυμάτων κάθε χρόνο, αλλά τα οποία είναι πιο περιοριστικά και ζουν σε δύσκολα κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια, το μεγαλύτερο μέρος των κέντρων αυτών, έχει μια πολυκλαδική αντιμετώπιση των θυμάτων βασανιστήριων, το οποίο σημαίνει ιατρική φροντίδα, ψυχολογική φροντίδα, κοινωνική ενσωμάτωση, ε, παροχές κινησιοθεραπείας, όλα αυτά. Θέλω να κάνω μια σύντομη παρουσίαση για τα θύματα βασανιστήριων στην Ευρώπη, να σας δείξω ποια είναι η κατάσταση. Ξέρετε ότι τα βασανιστήρια είναι ένα διεθνές πρόβλημα και εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η πρακτική σε πολλές χώρες της του κόσμου. Ένα 30% των ετούντων ασύλου υπολογίζεται ότι υπήρξαν θύματα ασύλου. Επομένως, από τα 2,9 εκατομμύρια που έχουν έρθει στην Ευρώπη θα είναι ένα σημαντικό ποσοστό το οποίο υπήρξε θύμα βασανιστήριων. Είναι μια ομάδα ευάλωτη ατών, ετών των ασύλου που αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας ψυχολογικής και σωματικής. Και αυτό είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τα θύματα, για τις οικογένειές τους αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας. Το δικαίωμα προς την υγεία, για την υγεία θεωρείται θεμελιώδης σε πολλούς ε, δημόσιους σε, πολλούς, ε, σε πολλά δημόσια και διεθνή έγγραφα. Υπάρχει λοιπόν ένα, ένα πρόβλημα να αντιμετωπιστούν τα άτομα αυτά και να υπάρξει η εποκατάσταση της ψυχολογικής και σωματικής τους υγείας. Αυτό πρέπει να είναι μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία χρηματοδοτεί αυτά τα ιδρύματα αποκατάσταση με τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το γεγονό ότι πάβει η χρηματοδότηση αυτού του Ιδρύματο σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσουν και πολλά τέτοια κέντρα αποκατάσταση. Για ορισμένα κέντρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χάσουν 60% τη χρηματοδότησή του από τη μια χρονιά στην άλλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα για μα. Το θέμα της αναγνώρισης των θυμάτων βασανιστήριων όπως είδαμε και σε αυτά που είπε ο κύριος Δεμποκέρ και οι προηγούμενοι ομιλητές, το θέμα της αναγνώρισης είναι θεμελιώδες. Όταν ξέρουμε ότι τα ευάλωτα αυτά θύματα θα πρέπει να ε, τύχουν θετικών μέτρων για την πρόσβαση σε περίθαλψη και σε σχέση με τις συγκεκριμένες ηλικέ συνθήκες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, το να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τα άτομα αυτά, αυτό είναι κάτι το κεφαλαιόδες για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα μέτρα προστασίας. Νομίζω ότι η αναγνώριση θα πρέπει να γίνει ως το δυνατόν πιο έγκαιρα για να εξασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα ακολουθηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες στα άτομα αυτά. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι να δημιουργηθεί μια ατομική μια πρώιμη ατομική αναγνώριση το ταχύτερο δυνατό στη διαδικασία αντιμετώπισης των αιτήσεων ασύλου για να εξασφαλιστεί η καλύτερη αντιμετώπιση των ετούντων αυτών ασύλου. Έχουν προσπαθήσει διάφοροι εταίροι μας να, ε, να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο το οποίο βοηθά ε, την αναγνώριση σε κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι δεν έχουν την κατάρτιση ως ιατροί, ως ψυχολόγοι για το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης των ε, ετούντων ασύλου. Τα πρώτα αποτελέσματα από αυτό το σχέδιο, το Protect, είναι θετικά και εμείς θα θέλαμε αυτή η διαδικασία αναγνώρισης να ενσωματωθεί στο γενικότερο σύστημα υποδοχής των ε, ε, ετούντων ασύλου. Έχω εδώ ένα φυλάδιο από το σχέδιο Protect. Μπορείτε να βρείτε και στην είσοδο της αίθουσας περαιτέρω φυλάδια και αν θέλετε περισσότερα αντίτυπα μπορείτε να απευθυνθείτε σε μένα. Μπορώ να σας φέρω την απαραίτητη τεκμηρίωση αν θέλετε. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της τεκμηρίωσης των περιπτώσεων βασανισμών ο στόχος της παρέμβασης επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και της ψυχικής υγείας δεν είναι μονάχα η αποκατάσταση, αλλά είναι απαραίτητος, η απαραίτητη αυτή η παρουσία τους για να τεκμηριωθούν τα βασανιστήρια τα οποία έχουν υποστεί. Δεν είναι μονάχα λοιπόν για την χορήγηση ασύλου, αλλά και για την έναρξη δικαστικών διαδικασιών κατά των βασανιστών, κάτι το οποίο το γνωρίζουμε πολλές φορές. Εδώ υπάρχουν πρότυπα όπως το πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης για να εξασφαλιστεί η ποιότητα της τεκμηρίωσης και να αποφύγουμε ότι αυτό το στάδιο της απόκτησης στοιχείων θα είναι επιπλέον τραυματισμός για τα άτομα που έχουν υποστεί βασανισμούς. Δυστυχώς αυτά τα πρότυπα δεν χρησιμοποιούνται πάντα. Για να κλείσω λοιπόν, τρεις ε, συστάσεις που απορρέουν από αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Προτείνουμε να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο θα έχει έγκαιρη, έγκαιρη αναγνώριση των ατόμων που έχουν αντιμετωπίσει τραυματικές συνθήκες βασιλανιστηρίων. Δεύτερον, να αναγνωριστεί με κατάλληλη φροντίδα και θεραπεία η κατάσταση αυτών των ατόμων. Και τρίτον, να υπάρξει και η παρουσία ιατροδικαστική ε, μέρημνα για να μπορέσει να υπάρξει τεκμηρίωση που θα οδηγήσει σε περαιτέρω διώξει. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι μια σαφέστατη παρουσίαση. Μας παρουσιάσατε όλες τις προκλήσεις ε, για τα θέματα πιθανών ε, προσφυγών και ξεπερνάμε λίγο και το θέμα του ασύλου σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε χρόνο για ένα-δύο πολύ σύντομες, πολύ σύντομες το επισημένο ερωτήσεις που ελπίζω να μην οδηγήσουν σε πολύ μακροσκελείς απαντήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από πλευράς μελών ή ήταν, αν ήταν όλα τόσο σαφή. Ο κύριος Μασί Πιντάλγο, ο οποίος άλλωστε όπως θα θυμάστε είναι και εισηγητής για τα θέματα της ε, κράτησης ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όλα όσα άκουσα από το πάνελ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι στον ε, εκπρόσωπο του Ιδρύματος για τους Βασανισμούς. Έχουμε τα ευάλωτα άτομα και τα, θέμα τα άτομα τα οποία είναι θύματα βασανιστήριων Υπάρχει κάποιος κατάλογος ε, ταυτοποίησης ε, όχι ανθρώπων αλλά χωρών στις οποίες ε, υπάρχουν πρακτικές βασανιστήριων. Διότι θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις εθνικές καταστάσεις για να μπορέσουμε να επισημάνουμε ποιες είναι οι χώρες οι, από, οι οποίες ακόμα εφαρμόζουν πρακτικές βασανιστήριων που οδηγούν σε ανθρώπους θύματα και θα θέλαμε να το γνωρίζουμε εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να σημειώνεται ότι αυτές οι χώρες εφαρμόζουν βασανιστήρια και να υπάρχουν και στις εκθέσεις της Διεθνούς Αδημιστίας, ώστε ε, να χρησιμοποιηθεί αυτό ως μέτρο ε, από πλευράς μας σε άλλους τομείς. Ευχαριστώ. Βεβαίως ότι συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέτε η καθημερινή μας προσπάθεια είναι ακριβώς ε, να προωθήσουμε τα ζητήματα αυτά. Αλλά ξέρετε, πολύ συχνά είναι δύσκολο να περάσουμε τα μηνύματα αυτά, γιατί ε, οι περισσότεροι δεν θέλουν τα βασανιστήρια ή δεν θέλουν να βλέπουν τα βασανιστήρια. Ε, επανειλημμένα εμείς και πολλά χρόνια είχαμε ε, καταγγείλει τις καταστάσεις την ισίων που ερχόντουσαν σε μας σαν θύματα βασανιστήριων, ενώ στη Γαλλία η κυρίαρχη άποψη ήταν ότι την ισιων είναι μια εξαίρετη χώρα και ακόμα πιο εξαίρετος τόπος διακοπών. Χρειαζόμαστε επομένω και μια ισχυρή πολιτική στήριξη έτσι ώστε να μεταφέρουμε αυτά τα ηχηρά μας μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αυτό ε, μας παραπέμπει και σε ένα άλλο θέμα το οποίο έθιξαν κάποιοι άλλοι, πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής ε, και λοιπά στοιχεία. Ε, έχουμε και τη σχετική έκθεση και το Ευρωπαϊκό Γραφείο υποστήριξη Ασύλου έχει αναλάβει αυτό το καθήκον. Και το πώς ε, θα απαντήσουμε βεβαίως καταλήλως, ε, όχι απλώς ε, μέσω μιας υπογραφή ενό μνημονίου συνεννόησης για να επιστρέφονται τα άτομα αυτά στις χώρε του. αλλά να λάβουμε και συγκεκριμένα μέτρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους ομιλητές του συγκεκριμένου τμήματος της συνεδρίασης τώρα. Μας δώσετε μια πολύ σαφή εικόνα πολύ πλούσια η οποία έχει προκύψει και από την εμπειρία σας. Στο επόμενο ε, τμήμα της συνεδρίασης ε, θα προεδρεύσει η συνάδελφος η Σεσίλια Βίπστρομ για το θέμα των ανηλίκων παιδιών και φαντάζομαι ότι θα είναι το ίδιο επικοδομητικό. Σεσίλια λοιπόν, έχεις τα ενία. Ελπίζω να είχατε ένα λεπτάκι να γνωριστείτε με κάποιους που δεν γνωρίζετε, έτσι. 30 δευτερόλεπτα ακόμα σας δίνω και μετά θα ξεκινήσουμε, διότι χρειάζεται λίγη περισσότερη ενέργεια εδώ. Γνωριστείτε μεταξύ σας, χαμογελάστε ο ένας τον άλλον. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο τρίτο τμήμα της συνεδρίασής μας. Ε, είμαι η Σεσίλια Βίκστρομ, είμαι από τη Σουηδία Ευρωβουλευτής από το 2009 και είμαι η συγγήτρια για το ε, θέμα της αναδιατύπωσης του Δουβλίνου 2. Ξέρουμε ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες ε, καταστάσεις και είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν τμήμα της συνεδρίασης ε, θα σταθούμε στα ανήλικα παιδιά που αναζητούν άσυλο και ξέρουμε φυσικά ότι τα ανήλικα παιδιά είναι ένα πολύ σημαντικό οριζόντιο ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει σε όλα τα ζητήματα ασύλου. κατά τη διάρκεια της ε, προετοιμασίας ε, της δέσμης των οδηγιών για το κοινό σύστημα ασύλου. Ε, σήμερα έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες στο ε, τμήμα αυτό της συνεδρίασης. Δεν θα σας καθυστερήσω εγώ και δεν θα σας ε, μιλήσω άλλο. Θα δώσω το λόγο στους ομιλητές για να μάθουμε τα θέματα από τους ειδικού. Καταρχάς λοιπόν η κυρία Ρεμπέκα Οντόνελ, η οποία είναι υπεύθυνη πολιτικής και ευαισθητοποίησης για άσυλο μετανάστευση στη Διεθνή Ένωση Save the Children από το 2007. Το Save the Children είναι μια παγκόσμια οργάνωση ανεξάρτητη για τα δικαιώματα των παιδιών και τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου των παιδιών αποτελούν μία από τις προτεραιότητές τους. Το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολείται με την νομοθεσία για το άσυλο και την εμπορία παιδιών την οδηγία για τις επιστροφές και το πρόγραμμα δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Επίσης, ε, ε, συνεργάστηκαν και με το πρόγραμμα για τα παιδιά τα οποία έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους ε, και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα ανά την Ευρώπη που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Με χαρά λοιπόν σας δίνω το λόγο κύριε Αντώνελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τα εισαγωγικά σας σχόλια και ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση να παραβρεθώ εδώ και να αναφερθώ στο θέμα των παιδιών στην νομοθεσία ασύλου και φυσικά τη θέση που μπορεί να λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Όπως είπε και η κυρία Βίκστρομ, παρακολουθήσαμε την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Ασύλου εδώ και αρκετά χρόνια και έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά τα παιδιά και για παιδιά σε οικογένειες που κάνουν αίτηση ασύλου, αλλά και παιδιά τα οποία μπορεί να ε, έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους και να ταξιδεύουν ασυνέοδευτα και να ζητούν άσυλο. Θα σταθώ λίγο στις βασικές μας θέσεις όσον αφορά τα παιδιά πριν ε, σταθώ στην κατάσταση των παιδιών ε, στις προτάσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή και στο τέλος θα επικεντρωθώ λίγο σε κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να απασχολήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εφαλτήριο ξεκινούμε από το γεγονός ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητα άτομα με συγκεκριμένα δικαιώματα και θα πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε ως παιδιά ανεξάρτητα από το καθεστώς μετανάστασης το οποίο βιώνουν. Εάν είναι ασυνόδευτα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους θα πρέπει να την χάνουν ειδική μεταχείριση και για να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση θα ήθελα να επισημάνω το εξή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι τα συνόδευτα παιδιά που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρε θα πρέπει να τίθενται υπό την ε, προστασία των ευρωπαϊκών κρατών ε, επιμονή μου βάσεως. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για κάθε ένα από τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες του ανάγκες κάθε φορά. Οι χώρες με είναι υποχρεωμένες και βάσει διεθνούς και βάσει ευρωπαϊκού δικαίου να εξετάσουν την κατάσταση του κάθε παιδιού και να καθορίσουν κατά πόσον ε, θα πρέπει να παραμείνουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες χώρες για το μέλλον. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να διέπεται από το συμφέρον τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες τους ανάγκες και φυσικά το γεγονός κατά, ε, πόσον είναι πρόσφυγες. Ε, αυτό βέβαια είναι κοινή λογική και κανονικά θα έπρεπε αυτό να είναι και ο χρυσός κανόνας σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βλέπουμε και στην οδηγία για την εμπορία και τις επιστροφές και είναι και προεξάρχον στοιχείο στο, στα προτινόμενα μέσα για το άσυλο. Είναι λοιπόν πολύ ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι ως αρχή ε, προβάλλεται όλο και περισσότερο στην νομοθεσία μας. Αλλά αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι ότι η αρχή αυτή για το βασικό συμφέρον των παιδιών δεν θα πρέπει να αντιγράφεται σε κάθε νομοθεσία και να θεωρείται ότι είναι μία αρχή η οποία εκτελείται αυτόματα ή και ότι τα κράτη-μέλη ε, μπορεί να λάβουν υπόψη την εφαρμογή της ε, απευθείας. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένε δικλείδε ώστε να υπάρχει και αρχή της αναλογικοτητας η οποία θα πορεύει από αυτή την αρχή υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που περιλαμβάνουν βασικές δικλείδες ασφαλείας, τι οποίες θα ήθελα να σταθώ τώρα. Καταρχά, να σα υπενθυμίσω ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία για το άφησιλο υπάρχουν μέτρα για τα συνόδευτα παιδιά, μέτρα για τι χωρισμένε οικογένειε, αλλά ουσιαστικά τα παιδιά είναι αόρατα. Δεν υπάρχει καν ορισμό του παιδιού ω άτομα κάτω των 18. Οι νέες διαπραγματεύσεις όμως ε, έχουν καλύτερες ε, δυνατότητες υποδοχής για τα παιδιά, καλύτερη οικογενειακή ζωή, βελτιωμένες πτυχές ε, ασούλου και μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν ότι θα εισακούονται τα παιδιά και θα γίνεται κατάλληλη αξιολόγηση. Και εμείς χαιρετίζουμε αυτή την πρόοδο, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης κάποιων διατάξεων και μας ανησυχεί το γεγονός ότι κάποιες από αυτές τις βελτιώσεις γίνονται υποπίεση στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ο στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πρόοδο στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα είναι σαφέστερε κάποιε διατάξει. Θα ήθελα να σας δώσω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα βελτιώσεων τα οποία ε, αποτελούν πρόκληση αυτή τη στιγμή και θα σταθώ και σε τρία σημεία τα οποία ίσως θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Καταρχάς, τα θα σας επλήξει είναι το θέμα της κράτησης και ξέρω ότι η κράτηση θα συζητηθεί ε, αργότερα πιο διεξοδικά. Στην πρώτη πρόταση αναδιατύπωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια διάτεξη για την κράτηση των ασυνόδευτων παιδιών και στη δεύτερη αναδιατύπωση ε, άλλαξε αυτό. Στη νέα πρόταση η κράτηση των ασυνόδευτων παιδιών μπορεί να γίνει αν είναι προς το συμφέρον τους. Ε, δύσκολα όμως μπορούμε να φανταστούμε πότε είναι προς το συμφέρον τους. Η ε, ενδείξεις ότι, υπάρχουν ενδείξεις ότι ε, υπάρχει χρήση ε, βίας κατά των παιδιών και νομίζω ότι το να, υποκράτη, να είναι παιδιά υποκράτηση εμένα μου φαίνεται μεσαιωνικός κανόνας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει το βάρος της απόδειξης ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους να κρατούνται τα παιδιά. Θεωρούμε γενικώς ως γενικό κανόνα ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να τελούν υποκράτηση. Υπάρχει και μια εκστρατεία του χρόνου ε, για να σταματήσει η κράτηση των παιδιών σε αυτές τις διαδικασίες και νομίζω ότι το υλικό για την εκστρατεία αυτή θα πρέπει να ενδιαφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης υπάρχει το θέμα της ενότητας της οικογένειας. Υπάρχουν ορισμοί για τα μέλη της οικογένειας στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά το Κοινοβούλιο τα έχει συζητήσει αυτά και όσον αφορά την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και εκεί στο Κοινοβούλιο υπήρχε ένας πιο περιοριστικός ορισμός για τα μέλη της οικογένειας από τον προορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην κάνει το ίδιο πράγμα για την οδηγία για την ε, υποδοχή παιδιών, αλλά θα πρέπει να υποστηρίξει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα ε, παιδί ε, που δεν συνοδεύεται από το, τη σύζυγο ή το σύζυγο θα πρέπει να θεωρείται ανάλογο. Τα παιδιά και τα παντρεμένα παιδιά είναι σοβαρό πρόβλημα. Τα παιδιά είναι παιδιά ανεξάρτητα από το αν είναι παντρεμένα ή όχι. Και υπάρχουν φυσικά και όλοι οι καταναγκαστικοί γάμοι. Ε, βρίσκονται λοιπόν σε συνθήκες ιδιαίτερα ευάλωτες και υπάρχουν ανάγκες προστασίας. Και θα θέλαμε και είναι προ όφελο των κρατών μελών να επιτρέπεται σε οικογένειε να μπορούν να επανενωθούν για να διωθεί και μια αίσθηση ασφάλεια. Και τώρα, εν συντομία, θα ήθελα να σταθώ σε τρεις διατάξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Καταρχάς, ε, οι κηδεμόνες. Οι κηδεμόνες που προσωπούν τα παιδιά είναι εκεί για να προστατεύσουν τα παιδιά και για να διασφαλίσουν ότι ε, λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των παιδιών. Δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε οργανισμός όμως πίσω από αυτούς που να, είναι, ε, να έχει συγκεκριμένα συμφέροντα. Παραδείγματο χάρη κάποιοι οι οποίοι ε, μπορεί να σχετίζονται ε, με την υπηρεσία συνόρων και μετανάστευση. Ε, αυτό το έλαβε υπόψη του το Κοινοβούλιο στην ε, ε, πρόταση για την υποδοχή μεταναστών και λέγεται ότι άτομα τα οποία έχουν ένομο συμφέρον και σχέση με άλλες υπηρεσίες δεν θα πρέπει να είναι κυδωμένες των παιδιών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχυθεί αυτή η ρήτρα και θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω ο κανόνας αυτός. Η αξιολόγηση τώρα της ηλικία. Αυτό είναι πάρα πολύ ακαθόδε ζήτημα, πολύ δύσκολο. Πώ μπορεί κάποιο να διαπιστώσει την πραγματική ηλικία ενός παιδιού. Χρειάζεται ένα μηχανισμό για να καθορίσουμε κατά πόσο ένα παιδί είναι όντως παιδί, ανήλικο παιδί. Και να τονίσω εδώ ότι δεν υπάρχει ακριβώς ε, διαδικασία διαπίστωσης της ηλικία ενός παιδιού. Θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα να υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να λαφθεί υπόψη πλήρω αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα επιτρέπεται ε, να ε, γίνεται συνεχώς έλεγχος με ακτίνες για να διαπιστωθεί η ηλικία ενός παιδιού. Τώρα, έχει υπάρξει κάποια πρόοδο για το κατά πόσον ένα συνόδευτο παιδί θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη χώρα βάσει του Δουβλίνου 2. Αλλά το Κοινοβούλιο εξετάζει περαιτέρω τα ζητήματα αυτά και κατά εμά θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που θα λαμβάνει υπόψη των συμφέρον των παιδιών, να συμπεριτέχουν ε, ε, οι βασικοί παράγοντε από κάθε χώρα και να υπάρχει κατάλληλη δυνατότητα φροντίδα ε, και εκειδαιμονία των παιδιών. Θα ήθελα να σας παρακινήσω να δείτε και την ιστοσελίδα μας για να δείτε τις θέσεις μας πιο αναλυτικά. Και τέλος, ε, πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να ε, αναφερθώ σε κάποια από τα βασικά επιχειρήματα που εμφανίζονται κατά των συγκεκριμένων διατάξεων. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ δαπανηρές και ότι δεν μπορούν να παράσχουν αποτελεσματική προστασία. Ε, Αυτά είναι επιχειρήματα τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του πολύ σοβαρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά κατά την άποψή μου αυτά τα πρακτικά επιχειρήματα δεν μπορούν ποτέ να είναι ει βάρον της υποχρέωσης της βασικής ανάγκης για δικλείδες ασφαλείας. Τα δικαστήρια το γνωρίζουν και πολλές φορές είναι υπόλογα τα κράτη-μέλη διότι δεν έλαβαν υπόψη τους το συμφέρον των παιδιών και για λόγους ουσίας αλλά και για διαδικαστικούς λόγους. Και η δεύτερη παρατηρήσή μου είναι ότι αυτές οι δικλείδες ασφαλείας δεν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολες και πολύ δαπανηρές στην εφαρμογή τους. Καταλαβαίνουμε ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν δίλημα και δεν ξέρουν ε, πώς ακριβώς να αξιολογήσουν και να βρουν ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού. Αλλά προσπαθούμε να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη ώστε να γίνεται αποτελεσματικά αυτό. Για παράδειγμα, συνεργαστήκαμε με το Φιλανδικό Υπουργείο για το πώς ε, παίρνουμε συνέντευξη από ένα παιδί ε, και ε, η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα κατάλογο θεμάτων τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη του ένα κράτος μέλος όταν επιστρέφεται ένα παιδί. Υπάρχουν λοιπόν και κατευθυντήριες γραμμές για το συμφέρον των παιδιών και όλα αυτά θα πρέπει να ενδιαφέρουν την όλη διαδικασία ασύλου. Είναι εδώ και το Νίντους και το ECI που ασχολούνται με τα θέματα των παιδιών και των ασυνόδευτων παιδιών και θεωρώ ότι όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη για να έχουμε αυτές τις δικλείδες ασφαλείας. Εν κατακλείδη να σας πω ότι θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ώστε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να δημιουργήσει ένα κατάλληλο πλαίσιο που θα προστατεύει τα ευάλωτα παιδιά στην πραγματικότητα και όχι μόνο στα χαρτιά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much πολύ. Προχωρούμε αμέσως δόκτωρα η οποία είναι διευθύντρια προγράμματος στη νομική έρευνα για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Βιέννη από το 2009 και είναι επικεφαλής τη για τα δικαιώματα των παιδιών στον Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Παρακαλώ προσπαθήστε να τηρήσετε το χρόνο που έχουμε ώστε κάποιοι να έχουν το χρόνο να θέσουν και κάποια ερωτήματα στο τέλος της, ε, της, της, ε, της παρουσίασης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παρουσίαση αυτή, την, την ε, παρουσία μας εδώ. Θέλω να παρουσιάσω την κατάσταση των παιδιών που είναι αποχωρισμένα από την οικογένειά τους. Έχετε εδώ αυτό το, τη δημοσίευση του φορέα μας σε σχέση με το θέμα αυτό η έκθεσή μας ακολουθεί μια προσέγγιση που έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Τα παιδιά τα οποία ήταν στην, ε, στην έρευνα αυτή συμμετέσχαν κυρίως μέσω συνεντεύξεων. Ήταν 336 παιδιά, 16 και πάνω στην ηλικία τους. Αντιμετωπίζει αυτή η έκθεση τις προστοκίες και τις απόψεις αυτών των παιδιών και των του προσωπικού που αντιμετωπίζει τα παιδιά. Αυτό είναι ένα τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι αποδεκτέ και επαρκεί οι πρακτικέ μα και αν χρειάζεται να τι αλλάξουμε και να έχουμε μια καλύτερη ενόραση στον τρόπο που βλέπουν τα παιδιά αυτή τη διαδικασία. Έχουμε λοιπόν ιδέες που ασχολούνται και με, το, με την ε, Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και θέλει να συμπληρώσει τη μελέτη του δικτύου για τις μεταναστεύσεις στην Ευρώπη σε σχέση με τις νομικές ρυθμίσεις για τους ανήλικους. Ήταν 12 χώρες οι οποίες ενεπλάξαν σε αυτή την έρευνα και τις έχετε στο, στο γράφημα αυτό. Αντιμετωπίζουμε στην έρευνά μας και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών που είναι η στέγαση, στέγαση η κοινωνική προστασία, η η περίθαλψη σε ιατρικό επίπεδο, η εκπαίδευση κτλ και αναψυχή και επίσης καλύπτει τα νομικά θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν τα παιδιά. Η κυδαιμονία, η εκπροσώπηση ενώπιον του νόμου, η καθορισμός του τι είναι παιδί, η ανείχνευση και η επανένωση των οικογενειών, τη διαδικασία ασύλου κτλ. Νομικές ε, νομικές πτυχές και διαδικασίες που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πρωταρχική σημασία στα παιδιά. Πολλές φορές όμως τα παιδιά δεν έχουν πληροφόρηση σε σχέση με τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες που τα εμπλέκουν. Πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έρευνες και οι ερωτήσεις προς τα παιδιά δεν είναι φιλικές προς τα παιδιά ή δεν έχουν ευαισθησία σε πολιτιστικό επίπεδο. Πολλές φορές δεν υπάρχει παρουσία νομικών συμβούλων και υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν και αποτελεσματική νομική βοήθεια στα θέματα αυτά. Η πτυχή της νομικής κυδαιμονίας. Αυτή θεωρήθηκε πάρα πολύ θετική, αλλά τα περισσότερα παιδιά δεν ήξεραν αν έχουν κάποιο κυδεμόνα ή ποιο είναι ο κυδεμόνα του ή ποιε είναι οι ευθύνε που έχει αυτό το άτομο. Σε ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι οι ενήλικες είναι οι κηδεμόνες, όταν αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Υπήρξαν καθυστερήσεις για τον καθορισμό ενός κηδεμόνα και υπήρξε έλλειψη απαραίτητης κατάρτισης και έλλειψη επαγγελματικής αντιμετώπισης στα θέματα αυτά. Ένα από τα παιδιά μου παιδιά που είναι, αναφέρεται στην έκθεσή μου, λέει δεν ξέρω τι είναι ο νομικός κηδεμόνας και δεν έχω κηδεμόνα για τον καθορισμό της ηλικία. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, μεταξύ των οποίων και χρήση τεκμηρίων. Αλλά τα ιατρικές δοκιμασίες πολλές φορές είναι συχνές και δεν υπάρχει, σε, δεν υπάρχει σαφήνεια σε σχέση με το είδος των τεστ, με την απαραίτητη πληροφόρηση για τα παιδιά, με το να υπάρξει συνένεση από τα παιδιά και για τους μηχανισμούς προσφυγής εναντίον τέτοιων καθορισμών ηλικίας. Για την ανείχνευση των οικογενειών και την επανένωση. Τα περισσότερα παιδιά θέλουν να επανέλθουν στον οικογενειακό τους χώρο, αλλά πολλές φορές δεν υπάρχει πληροφορία για την ανέχνευση αυτών των οικογενειών, δεν υπάρχει επιτυχία στη διαδικασία για την ε, ανείχνευση των οικογενειών. Δεν υπάρχει βοήθεια από το Διεθνή Σταυρό, Ερθρό Σταυρό και τις ε, που να είναι πάντα αποτελεσματική και περιορισμένα παιδιά δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις διαδικασίες και δεν θεωρούν ότι θα βοηθήσει την αίτηση ασύλου τους. Για την διαδικασία ασύλου. Τα παιδιά θέλαν πράγματι να συζητήσουν αυτή τη διαδικασία στις περισσότερες χώρες, αλλά η διάρκεια της διαδικασίας για την αναγνώριση του νομικού καθεστώτος τους οδηγεί σε αβεβαιότητα. Τα παιδιά πολύ συχνά δεν έχουν πληροφορίες σε σχέση με το ρόλο των εμπλεκομένων στη διαδικασία ασύλου δεμόνες και σύμβολοι κτλ. Πολλά παιδιά νιώθουν ματέωση γιατί δεν έχουν αρκετό χρόνο να συζητήσουν την περίπτωσή τους με τους νομικούς συμβούλου και δεν υπάρχουν πάντα οι κατάλληλοι διερμηνεί ή αυτοί που γνωρίζουν τη γλώσσα και τη διάλεκτο που μιλούν τα παιδιά και πολλές φορές υπάρχει και πρόβλημα μεροληψίας από την πλευρά των διερμηνέων. Κράτηση. Πολύ λίγα παιδιά έχουν ε, τύχει συνέντευξη κατά τη διάρκεια τη κράτηση, αλλά όλοι μιλήσαν, όλα τα παιδιά μιλήσαν για τι εμπειρίε του. Δεν είναι εύκολο τα παιδιά να καταλάβουν γιατί τα κλειδώνουν, αν δεν έχουν κάνει κάποιο αδίκημα. Σε ορισμένα τα παιδιά κρατούνται συστηματικά από τη στιγμή που φτάνουν μέχρι να καθοριστεί η ηλικία του. Σε ορισμένε περιπτώσει αναφέρθηκαν ότι δεν υπήρξε καμία μορφή νομική βοήθεια κατά τη διάρκεια τη κράτηση. Σε ορισμένα είπαν τα παιδιά ότι υπέστησαν σωματική και ψυχολογική βία κατά τη διάρκεια της κράτησης. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα αναφερθώ μονάχα σε ορισμένε πτυχέ για τι συνθήκε εργασία των παιδιών. Για την στέγαση. Θετικό είναι το γεγονό ότι ήταν μικρότερη η κλίμακα στέγαση και όχι μαζική στέγαση. Αυτόνομη ή αυτόνομη στέγαση για τα παιδιά άνω των 16. Από την αρνητική πλευρά Πολλές φορές τα παιδιά τίθενται σε κέντρα κράτησης, σε ξενοδοχεία ή σε πανδοχεία και πολλές φορές στεγάζονται μαζί με άσχετους ενήλικες. Και υπάρχουν προβλήματα συμφόρησης και υπερβολικού αριθμού στεγαζόμενων σε ορισμένε περιπτώσεις. Τα παιδιά προτιμούν να ζουν σε μεγαλύτερες αστικές περιοχές, ενώ οι ενήλικες είχαν διαφορετικές απόψεις. Αυτό έχει να κάνει με την ε, μέρημνά τους και την ασφάλεια των παιδιών. Τα κέντρα αρχικής υποδοχής θεωρήθηκαν ότι παρέχουν μη επαρκείς συνθήκες διαφύωσης σε σχέση με την πρόσβαση σε, ε, σε περίθαλψη, πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα, ιδιωτικότητα, παροχή τροφίμων κτλ. Για την υγειονομική περίθαλψη, τα περισσότερα παιδιά είχαν θετικέ εμπειρίε, αλλά υπήρξαν και προβλήματα έλλειψη ε, ιατρικού ελέγχου όταν έφταναν στα κέντρα αυτά, περιπτώσεις που δεν υπήρξε δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης. Η διερμηνία δεν ήταν πάντα επαρκής και κάποια κορίτσια είπαν προτιμούσαν γυναίκες ιατρούς, αλλά αυτό δεν ήταν πάντα δυνατόν. Παιδεία. Στα περισσότερα κατημέρια γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν στο κύριο ρεύμα τη παιδεία τα παιδιά αυτά, αλλά για τα παιδιά που βρίσκονται σε μεγάλα κέντρα στέγαση αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχουν δυσκολίε για την ένταξη στο σχολικό περιβάλλον. Σε ορισμένα κέντρα ε, υποδοχή η παιδεία είναι μονάχα γλωσσικά μαθήματα και τα παιδιά χρειάζονται περισσότερε ώρε εκπαίδευση. Ορισμένοι ενήλικε έχουν εκφράσει ανησυχίε για την πρόσβαση στο σχολείο και δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες φιλικές προς τα παιδιά για τις επιλογές σε σχέση με το σχολείο. Διακρίσεις και κακομεταχείρισεις. Η έρευνα δεν είχε σαν στόχο να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα και λίγα παιδιά αναφέρθηκαν σε αυτά. Αλλά έχουν αναφερθεί περιπτώσει καταχρηστική και βίαιη συμπεριφορά από την αστυνομία και άλλε αρχέ. Τα παιδιά πολλέ φορέ είναι υποχρεωμένα να επαναλαμβάνουν τι λεπτομέρειε τραυματικών εμπειριών του για να ελεγχθεί η ακρίβειά του. Νιώθουν προσβολή τα παιδιά που δεν του παίρνουν στα σοβαρά ή πολλέ φορέ του κατηγορούν για ότι λένε ψέματα. Υπάρχουν περιορισμένε δυνατότητε προσφυγή για τα παιδιά σε σχέση με την έλλειψη πληροφοριών για τα θέματα αυτά. Για να κλείσω, θέλω να πω ότι οι εμπειρίε των παιδιών αυτών ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσής τους και τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Οι απόψεις αυτές δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση των παιδιών και για τις ανάγκες τους. Και πολλές φορές αυτό γίνεται με μικρό κόστος και προσπάθεια. Και θέλω να τονίσω ότι το πρόγραμμα της Στοχόλμης που ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη τα ασυνόδευτα παιδιά να τύχουν ιδιαίτερης προστασίας και αντιμετώπισης και τονίζει ότι η ενίσχυση των τελωνιακών ελέγχων δεν θα πρέπει να εμποδίσει την προστασία για τα άτομα αυτά τα οποία πρέπει να υποφεληθούν από αυτήν. Ευχαριστώ. I thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δόκτωρα Μαρτίνε Τεμπάνες. θυμάμαι την ε, ε, συνάντηση που είχαμε τη συζήτηση με ένα 15χρονο Αφγανό ε, που ρωτούσε «Έχω δικαιώματα» Αυτό είναι ένα καλά κρατημένο μυστικό. και το μόνο που ήθελε ήταν να πάρει τηλέφωνο τη μητέρα του. Ήθελε να μιλήσει με τη μητέρα του. Αυτή είναι η κατάσταση για ένα 15χρονο ανήλικο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φερστέχεν, ο οποίος είναι διευθυντής του Νίντος γραφείο υποδοχής για συνόδευτα ανήλικα ε, παιδιά που αιτούνται ασύλο στην Ολλανδία. Η Νίντος είναι ε, υπεύθυνη για περίπου 300 συνόδευτα παιδιά. Εσείς αναλάβατε και την πρωτοβουλία δικτύωσης ε, των ε, αντιστοίχων γραφείων για συνόδευτα ανήλικα παιδιά και πλέον έχετε συνδεθεί με την Ιρλανδία, με τη Σουηδία και με άλλες χώρες. Με μεγάλη χαρά λοιπόν σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, που μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να συζητήσω την κατάσταση των ασυνόδευτων ανήλικων ε, παιδιών που ετούνται άσυλο. Έχουμε πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας ε, των ασυνόδευτων ανηλίκων και επομένως μπορώ να σας πω ότι το θέμα ανεξάρτητης κυδαιμονίας είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα ευάλωτα παιδιά. Ε, τα συστήματα κυδενομίας ε, ε, εκφαίνονται τελείως διαφορετικά από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και ε, χρειάζεται συνέργεια ανάμεσα και στα, στις υπηρεσίες ε, και τα Υπουργεία. Βεβαίως θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι αλλάζει η κατάσταση σύμφωνα με το πώς έχει μπει κανείς στην χώρα. Δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα κυδαιμονίας που, θα, που αφορούν και αναφέρονται στις ίδιες ε, υποχρεώσεις. Ε, δεν δημιουργούν δηλαδή, παρότι αναφέρονται σε διάφορες ε, περιπτώσεις, δεν αποτελούν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών αυτών. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση. Η υποχρέωση και η λογοδοσία θα πρέπει επίσης να καθοριστούν. Σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση η οποία θα έχει την σαφή ευθύνη ε, για να ξεχωρίζει τα παιδιά και θα πρέπει να είναι υπόλογοι για την ε, ευθύνη αυτή. Βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχουν και οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι, καθώς επίσης και σαφής εντολή για αυτή την οργάνωση η υπηρεσία. Θα σας δώσω ε, δύο παραδείγματα πολύ άσχημων ε, καταστάσεων όπου η οργάνωσή μας η ΝΙΤΟ ε, είχε και εξακολουθεί να έχει κεντρικό ρόλο έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι η δράση η οποία θα ληφθεί θα είναι η καλύτερη για το παιδιό. Η μία κατάσταση αφορά την επανένωση ενός μωρού που ζει στην Ολλανδία με τους παππούδες του που ζουν σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η άλλη κατάσταση αφορά ένα κορίτσι το οποίο ε, έχει κάνει προσφυγή βάσει του Δουβλίνου και έπρεπε να επιστρέψει σε μια άλλη χώρα της σύνθηκης του, Λονδίνου, ε, του Δουβλίνου όπου δεν είχε κανέναν ε, εκπρόσωπο της οικογένειάς του. Ε, καταλαβαίνουμε από τα δύο αυτά παραδείγματα ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν οι δομές αυτές οι οποίες θα διευκολύνουν την δράση η οποία θα είναι ε, καλές για το παιδί. Η πρώτη ε, περίπτωση αφορά την ε, μια κοπέλα 17 χρονών που έφτασε το 2008 όταν ήταν 14 για πρώτη φορά στην Ευρώπη από την ε, Λιβύη ενώ ε, προέρχεται από την ε, Ερυθρέα. Πρώτα απ' όλα από την Λιβύη έφτασε σε ένα στρατόπεδο προσφύγων σε μια χώρα, σε μια πόλη συγγνώμη, που έμεινε 8 μήνες. Εκεί είχε κάποια στήριξη από ομοεθνείς ε, Μετά όμως όταν έκλεισε αυτό το στρατόπεδο προσφύγων ε, ε, έμεινε στους δρόμους όπου στην ουσία έκανε, ζητούσε ελεημοσύνη και αυτό συντήθηκε σε ένα μήνα και μια οικογένεια από την Ερυθρέα τελικά την βοήθησε να φτάσει μέχρι την Ολλανδία. Τον Ιούνιο του 2009 λοιπόν η έρω έφτασε στην ε, Ολλανδία και ζήτησε άσυλο. Τον Ιούλιο του 2009 όταν ήταν πλέον 15 χρονών ε, ε, της δόθηκε η κυδαιμονία υπό την οργάνωση Νίντος. Η αίτησή της όμως απερίφθη γιατί είχε πρώτερα ζήσει σε μια άλλη χώρα της συμφωνίας του Δουβλίνου με αποτέλεσμα ε, έγινε αυτό που λέμε υπόλογη της ε, πρώτης ένταξης στην συνθήκη του Δουβλίνου και το Σεπτέμβριο του 2010 ε, τελικά κρατήθηκε έτσι ώστε να μετατοπιστεί σε άλλη χώρα παρότι η οργάνωσή μας η Νίντος ήταν σαφώς αντίθετη στην κατάσταση αυτή. Εν πάση περιπτώσει ε, καταλαβαίνετε ότι τελικά η Νίτος κατάφερε να κάνει κάποιες ε, διευθετήσεις ε, με άλλες ε, οργανώσεις και τέλος πάντων να συνεχίσει η κυδαιμονία της σε άλλες χώρες. Ε, όταν έφτασε στην ε, άλλη ε, χώρα, έφτασε, μπήκε στην φυλακή και μετά από λίγο διάστημα την αφήσανε στους δρόμους. Έζησε στους δρόμους, δεν είχε, στους πέντε δρόμους, κάτω από γέφυρες κοιμότανε, δεν είχε φαγητό, φοβότανε να ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία και στο τέλος αποφάσισε να επιστρέψει στην Ολλανδία. Η Νίντος ε, ήταν πεπισμένη της, ε, ότι έλεγε αλήθεια, ε, αποφάσισε να φέρει την ιστορία αυτή εις γνώση του αρμόδιου Υπουργείου. Δεν είναι βεβαίως η συνήθις διαδικασία και χρησιμοποιήθηκε από την Νίντο μονάχα κατ' για αυτήν την τόσο δύσκολη περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, μονάχα θυμάται τις φρικτές της εμπειρίες σε αυτή τη χώρα τη συμφωνία του Δουβλίνου και τρελαίνεται πραγματικά. Ε, είπε στους εκπροσώπους της Νίντος ε, ότι όλη η ζωή της τελικά ήταν περιπλάνηση και μιζέρια. Η Νίντος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να της ε, παράσχει ψυχοκοινωνική βοήθεια γιατί είναι απαραίτητη. Αλλά ακόμα δεν είναι καν σε θέση να δεχτεί τη βοήθεια αυτή. Η άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση του μωρού που ανέφερθηκα προηγουμένω. Είναι το μωρό που λέγεται Φεϊζή. Το μωρό Φεϊζή λοιπόν γεννήθηκε στο Ιράν ε, από Αφγανή μητέρα η οποία, ε, ε, η οποία κατέληξε στο Ιράν μαζί με αυτό το μωρό και την αδελφή του οι γονείς της ε, μητέρας ε, ζουν στην Βρετανία και έχουν βρετανική υπηκότητα. Λόγω της κατάστασης ε, και λόγω του προβληματισμού των γονιών για την κόρη τους και για τα εγγόνια τους, ταξίδεψαν στο Ιράν και προσπάθησαν να επιστρέψουν μαζί με την κόρη τους και με τα εγγόνια τους στην Βρετανία. Η μητέρα και τα παιδιά όμως είχαν ψεύτικα διαβατήρια και στο Ντουμπάι η μητέρα του Φεϊζή και οι αδερφοί του ε, συνελήφθησαν και ε, μάλλον θα εκτοπιστούν προς το Αφγανιστάν. Οι ε, παππούδες έφυγαν με τον Φέιζι και κατάφεραν να πάρουν την επόμενη πτήση για το Άμστερνταμ. Μόλις έφτασαν στην Ολλανδία, βεβαίως έγινε σαφές στον έλεγχο των διαβατηρίων ότι δεν υπήρχαν τα σωστά έγγραφα και ότι ο Φέιζι είχε ψεύτικο διαβατήριο οι, οι παππούδες παραδέχτηκαν ότι όντως ήταν ψεύτικα, ήταν πλαστά, το, πλαστό το διαβατήριο του Φέιζη. Ε, καταρχάς τους υποψιάστηκαν για εμπόριο βρεφών, αλλά τελικά επέτρεψε, τους τους ε, να συνεχίσουν το ταξίδι τους μέχρι την Αγγλία. Από τη στιγμή της σύλληψης ε, αναμίχθηκε η Νίντος με το θέμα αυτό και ε, ορίστηκε ως κηδεμόνας η Νίντος του Μωρού βάσει του δικαστηρίου των ε, ανηλίκων. Και βεβαίως οι προσπάθειες τη Νίντος εστιάστηκαν στην επανένωση του Φεϊζή με τη μητέρα του και με την αδερφή του. Η μητέρα από τηλεφώνου συμφώνησε με αυτήν την ε, επανένωση, ε, δηλαδή το να σταλεί ο Φεϊζή στους ε, παππούδες γιατί θεωρούσε ότι η επανένωση, η επανασύνδεση του μωρού με αυτήν θα ήταν ε, ανασφαλής για τον Φέιζη. Η Νίδος λοιπόν προσέγγισε όλες τις πιθανές υπηρεσίες και οργανισμούς όπως ας πούμε ε, την πρεσβεία των ε, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το γραφείο μεταναστών, ε, και τα ε, και το Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι ώστε να προσπαθήσει να προχωρήσει με την επανένωση της οικογένειας, αλλά τίποτα δεν έγινε. Η Κεντρική Αρχή επίσης ε, ετέθη εν γνώση του θέματος, αλλά τελικά απεφάνθη ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα η επανένωση του Φεϊζή με τους, ε, τους του στη Βρετανία. Ε, η μόνη λύση που μπορούσε να αντιμετωπίσει η Νίντος ήταν η αναχώρηση προς τη Βρετανία μέσω της διαδικασίας του Δουβλίνου. Ε, ζητήθηκαν αποσαφηνήσεις ε, έτσι ώστε να αποφασιστεί εάν θα ακολουθεί το τελικά η διαδικασία του Δουβλίνου και απεφασίστη να ζητηθεί από τις Βρετανικές Αρχές μέσω της διαδικασίας του Δουβλίνου να αποδεχθούν τον Φεϊζή. Ε, όμως ε, ε, παρότι η Νίντος μάζεψε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα υπέβαλε στις Βρετανικές αρχές, φάνηκε ότι δεν ήταν αρκετά και δεν επίστησαν. Επομένως αναγκάστηκε η Νίντος να κάνει ακόμα και εξέταση του DNA. Και βεβαίως εντωμεταξύ η Νίντος ήταν σε διαρκή επικοινωνία με, το δικαστήριο ε, ανηλίκων έτσι ώστε να υπάρξει ετοιμιγορία του δικαστηρίου ε, και να συνεχιστούν οι προσπάθειες ε, και να εξακολουθήσει και η στήριξη του Φεϊζή μετά από την επανένωση με τους, γονι με τους παππούδες του. Ε, οι επαφές ήταν πάρα πολύ δύσκολες ε, και τελικά ε, η τελική απόφαση του δικαστηρίου ανηλίκων της Ολλανδίας απεφάνθη ότι μπορεί να μετατεθεί η κυδαιμονία του παιδιού προς τους παπούδες. Εν πάση περιπτώσει, ο Φεϊζή βρίσκεται, βρέθηκε εντωμεταξύ μεταξύ για 11 μήνες στην Ολλανδία ε, και τώρα είναι 18 μηνών. Αυτή τη στιγμή η Νίντος ε, προσπαθεί να αντιμετωπίσει και τα, τις, ε, τα επιπλέον αιτήματα των Βρετανικών αρχών. Ε, όμως είναι σαφές ότι ο Φεϊζή δεν μπορεί να μείνει, πολύ με αυτήν την ε, οικογένεια με την οποία βρίσκεται τώρα, γιατί ε, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο ο αποχωρισμός από αυτή την οικογένεια όταν θα επανενωθεί με την δική του ε, οικογένεια. Και επομένω, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό άλλωστε σας ε, ε, μίλησα για, αυτά τα δύο, για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κηδεμόνας ο οποίος πραγματικά να ενδιαφέρεται για το παιδί και δεν είναι δυνατόν να κρατάμε μωρά ή με παιδιά 14 χρονών στην αγωνία και στην, στη μιζέρια. Αυτό είναι πραγματικά τελικά μιζέρια για την ίδια μας την κοινωνία. Επομένως ε, ε, ζητώ να μην συμπιέζονται τα δικαιώματα των μωρών και των ε, ανηλίκων παιδιών από τους γραφειοκράτες αυτού του πύργου της ε, Ευρώπης. Ε, θα πρέπει να βλέπουμε τις ε, περιπτώσεις με ανθρώπινο μάτι και επομένως να μην ξεπερνούν τους τρεις μήνες οι διαδικασίες από πλευράς των μεταναστευτικών αρχών έτσι ώστε, για, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Επίσης ζητούμε να διευθετήσετε το ζήτημα έτσι ώστε στην περίπτωση των προσφυγών ε, βάσει του ε, Δουβλίνου το παιδί να μπορεί ε, να μεταφερθεί από έναν κηδεμόνα σε έναν άλλον κηδεμόνα. Να μην αφήνεται δηλαδή στην τύχη του. Ε, θα θέλαμε ε, επίσης να βρούμε εταίρους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνουμε μια έκκληση και από αυτό το βήμα. Ε, αυτό σημαίνει οργανώσεις με τις οποίες μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή όταν έχουμε μια περίπτωση την οποία θεωρούμε πρωταρχικής σημασίας έτσι ώστε να βρίσκουμε λύσεις όταν ένας ασυνόδευτος, ένα ασυνόδευτο ανήλικο παιδί βρίσκεται σε μια ξένη συγκεκριμένη χώρα. Ε, νομίζουμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια καλή, ένας καλός ορισμός για την οικειδαιμονία και να εφαρμόζεται από όλους. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Όπως βλέπετε ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα. Σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε με το πρώτο τμήμα της συνεδρίασης ε, που καθυστέρησε περίπου μισή ώρα από την ώρα που είχε στη διάθεσή του και εδώ ε, έχουμε καθυστερήσει πολύ. Δεν θα ε, δώσω λοιπόν το λόγο για ερωτήσεις. Η Γραμματεία συμφώνησε να ε, συγκεντρώσει τις ερωτήσεις σας και να τις υποβάλουμε γραπτό στους εμπειρογνώμονες και να λάβετε επίσης και γραπτή απάντηση. Ολοκληρώνουμε λοιπόν λέγοντας ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το συμφέρον των παιδιών κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του κοινού συστήματος εσύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα η κράτηση δεν είναι κάτι το οποίο είναι ε, σύ, σύνομο με την Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που έχει αντίθετη άποψη, αλλά δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς να το αναφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια στη σημερινή ημέρα και θα πρέπει να συνεχίσουμε όλοι να προχωρούμε χέρι-χέρι. Γνωρίζουμε όλοι ποιο είναι ο δρόμος και όλους μας πιέζει η ίδια προθεσμία, το τέλος του 2012. Σας ευχαριστώ πολύ. of not Ελοχεύει ο κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μη συμμορφούνται προ το διεθνώ δίκαιο, προ τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα, καθώ επίση και προ την ομοθεσία του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Mm. Κυρίε και κύριοι, Σήμερα θα μπορούσα να μιλήσω για τις έννοιες των ασφαλών χωρών, ένα από τα αγαπημένα μου ζητήματα αλλά πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ούτως ή άλλως έχει συζητήσει αναλυτικά και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Θα μπορούσα να μιλήσω επίσης και για τις περίπλοκες διαδικασίες οι οποίες προκύπτουν ε, συνεπία πολλαπλών αιτήσεων. Θα μπορούσα κάλλιστα να απαντήσω σε ερωτήσεις αργότερα αν δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά επειδή ακριβώς μας πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα να σας δώσω μια εικόνα ε, για μία από τις προτάσεις ε, οι οποίες ε, παρουσιάζονται στην αναδιατύπωση. Την ε, βασική αρχή της έγκαιρης αντιμετώπισης, του front-loading. Τι σημαίνει η έγκαιρη αντιμετώπιση. Να το καταφέρουμε σωστά από την αρχή. Σημαίνει να έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να λάβουμε απόφαση πριν ή στην αρχή μιας διαδικασίας. Front loading σημαίνει να δημιουργήσουμε μια διαδικασία που θα μας επιτρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις ποιότητας στην πρώτη χρονική στιγμή ε, πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Διαδικασίες οι οποίες ε, επιβεβαιώνονται στη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο, ε, αποφάσεις οι οποίες δεν ακυρώνονται στη συνέχεια από το δικαστήριο. Η ποιότητα είναι ένας στόχος ο οποίος χρησιμοποιείται για να καθορίσουμε ποιες είναι οι καλές αποφάσεις, οι οποίες βάσει των καθορισμένων διαδικασιών αναγνωρίζουν αν υπάρχει κίνδυνος δίωξης και να χρησιμοποιηθεί ως σοβαρό όπλο στη χώρα ε, καταγωγής. Είτε αυτή είναι η Σομαλία, είτε είναι το Ιράκ, είτε οποιαδήποτε άλλη. Μία απόφαση ποιότητας είναι μία απόφαση η οποία δημιουργεί εκ των προτέρων Ποιο είναι πρόσφυγας και ποιο δεν είναι. Και είναι μια απόφαση η οποία σώζει ζωή. Ε, μια απόφαση η οποία καθορίζει ποιο χρειάζεται διεθνή προστασία και ποιο αντίθετα προσπαθεί να ε, εκμεταλλευτεί το σύστημα. Μία απόφαση ποιότητας είναι μία απόφαση που μας επιτρέπει να βρούμε τη σωστή λύση την πρώτη χρονική στιγμή. Το front loading είναι πλεονέκτημα για όσους κάνουν αιτήσει ασύλου. Και οι αιτήσει αυτές θα πρέπει να αναλύονται προσεκτικά σε εύλογο χρονικό διάστημα και δεν θα υπάρχει αβεβαιότητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα βρεθούν άνθρωποι να περιμένουν να ακούσουν τη μοίρα τους. Αλλά είναι και πλεονέκτημα για τα κράτη-μέλη, διότι θα μειώσει το κόστος το οποίο σχετίζεται με την ε, παροχή υλικού, συνθήκων ε, υποδοχής, ε, μικρότερο χρόνο για να λαμβάνουμε αποφάσεις και αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες υποδοχής, δηλαδή διατροφή, στέγαση και ρουχισμός, θα πρέπει να παρέχονται για συντομότερο χρονικό διάστημα και αυτό προφανώς θα μας οδηγήσει σε αποταμίευση, σε μείωση κόστους. Αν λάβουμε υπόψη όλα τα σωστά στοιχεία, αυτά θα επιβεβαιωθούν σε επόμενο στάδιο και αν φτάσουμε στο δικαστήριο μπορεί να οδηγηθούμε σε απόφαση να απορριφθεί η αίτηση εάν δεν είναι σωστή η απόφασή μας στην αρχή. Εξετάστηκε επίσης Τι επίπτωση έχουν ε, οι ε, διαδικασίες ετήσιων ασύλου στα κράτη-μέλη βάσει μιας μελέτης την οποία μπορείτε να βρείτε στην ε, τεκμηρίωση που σας δίνεται στην είσοδο. Στην έρευνα αυτή έχουμε 700 σελίδες αποδείξεων. Σε κάποια από τα κράτη-μέλη τα οποία αποτέλεσαν το κείμενο της έρευνας περίπου το 20% του συνολικού αριθμού των ανθρώπων που τη χάνουν καθεστώτος ε, διεθνούς προστασίας αρχικώς είχαν αρνητική απόφαση η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε από το δικαστήριο και έγινε θετική ε, το να υπάρχει άρνηση σε πρώτο στάδιο έχει διαφορετικές συνέπειες. Πολλοί ε, από τους ετούντες σε άσυλο ε, είναι αποθαρρυμένοι και δεν κάνουν έφεση. Δεν θα έκανε κάποιος έφεση αν ήξερε ότι υπάρχει 20% ποσοστό επιτυχίας. Εγώ θα έκανα. Οι διαδικασίες έφεσης είναι δαπανηρές. Ε, πολλές φορές θα πρέπει να δοθεί επιπλέον υλικό επιβίωσης, ηματισμός, ρουχισμός, όλα αυτά ε, αλλά ε, υπάρχουν συνέπειες και για την ίδια την απόφαση. Αν έχουμε λοιπόν έγκαιρη αντιμετώπιση, οι αρνητικές αποφάσεις θα επιβεβαιώνονται σε δεύτερο στάδιο αν έχουν ληφθεί σου καταλήλως και αποτρέπονται οι ε, εφέσεις και έτσι δεν θα υπάρχει επιπλέον κόστος για τις χώρες μέλη. Αυτό σημαίνει front loading. Να τα καταφέρουμε την πρώτη φορά <laughs> και να γλιτώσουμε χρήματα. Υπάρχει όφελος λοιπόν αν ε, υιοθετήσουμε αυτή τη διαδικασία της αναδιατύπωσης ε, και δεν θα υπάρχει κατάχρηση γιατί θα τους ε, εντοπίζουμε αμέσως. Τώρα, είναι μαγική αυτή η πρόταση. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις που μπορούν να συνεισφέρουν. Υπάρχουν διατάξεις για την επιμόρφωση και την κατάρτιση των αρμοδίων αρχών, διατάξεις για τις ε, πληροφορίες και για τις νομικές και τις διαδικαστικές πληροφορίες. Βελτιωμένη εμπειρογνωμοσύνη και επιπλέον πληροφορίες οι οποίες θα παρέχονται σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις ε, και πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής η οποία θα δίνονται από το Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου, το ΕΑΣΟ θέματα που αφορούν ε, μητρώα, ε, ε ιατρικά αρχεία και ούτω καθεξής. Να δούμε καταρχάς ε, τα στοιχεία ένα προς ένα. Η κατάρτιση και η επιμόρφωση του κατάλληλου προσωπικού. Εάν είναι κατάλληλα καταρτισμένο, μπορεί γρήγορα να βρει ποιος πράγματι χρειάζεται διεθνή προστασία και ποιος προσπαθεί να καταχραστεί το σύστημα. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι πολύ σημαντική για να έχουμε τη σωστή λύση την πρώτη στιγμή. Και αυτό φυσικά μπορεί να σας φαίνεται προφανές, αλλά στην έρευνα που σας ανέφερα προηγουμένως, διαπιστώθηκε ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη που αναλύσαμε, δεν απαιτούνται συνεντεύξεις για Ε, να είναι κάποιος υπεύθυνο για θέματα ασύλου και να ε, αποφασίζει ποιος είναι ε, ποιος επιλέγεται για διεθνή προστασία. Κάποιοι δεν έχουν καν προηγούμενη εκπαίδευση και τρία κράτη-μέλη δεν παρέχουν καμία εκπαίδευση σε κανένα επίπεδο πριν από την πρόσληψη. Καταλαβαίνετε λοιπόν πολύ εύκολα ότι η απέτηση εκπαίδευσης ε, μιας αρμόδιας αρχής για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στη διαδικασία ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες. Τον Ιανουάριο του 2012 το ΕΑΣΟ, το Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου, θα αναλάβει τα θέματα ευρωπαϊκού ασύλου. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα μας βοηθήσει να έχουμε πρακτική συνεργασία και χρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγος. Κατά την άποψή μας είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένες και να περιλαμβάνουν και αυτό τη βιβλιογραφία για το Ευρωπαϊκό Άσυλο. Επίσης, θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες για την ε, ρητή αλλά και έμεση απόσυρση μιας αίτησης. Αυτό θα μας βοηθήσει να μειώσουμε πολύ σημαντικά τον αριθμό των ε, πολλαπλών αιτήσεων που είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσα να συνεχίσω με τα ωφέλη του front-loading τις έγκαιρη αυτή αντιμετώπιση και τις διάφορες πτυχές, αλλά ξέρω ότι με πιέζει ο χρόνο. και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών τη να υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατόν ε, τα μέτρα για το άσυλο, και τις οδηγίες για τις κοινέ διαδικασίες για το καθεστώς διεθνούς προστασίας, το οποίο θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να τα καταφέρουν από την αρχή, να σώσουν ζωές και να εξοικονομήσουν χρήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα και ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέροντα τα λόγια σας. Θα δώσω το λόγο στην Άσο η οποία εκπροσωπεί το τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το 2010 είχε συμμετάσχει σε μια μελέτη για μια άλλη πτυχή του θέματος αυτού που είναι το δικαίωμα, η υποχρέωση πληροφόρησης σε σχέση με τις διαδικασίες των ετούντων ασύλου. Και αν θέλετε μπορείτε να μείνετε μέσα σε ένα χρονικό λογικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω από τη δική μου πλευρά για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση που απευθύνθηκε στο Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την έγκαιρη αντιμετώπιση. Θέλω να εστιάσω την προσοχή μου σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το φθινόπωρο έγινε το φθινοπόρο του 2010. Αφορά την πρόσβαση σε ουσιαστική, σε αποτελεσματική προσφυγή και την ανάγκη να πληροφορήσουμε τους ε, τούντες για τις διαδικασίες. Και εδώ εμπιπτεί το θέμα της έγκαιρης αντιμετώπισης. Το ερώτημα είναι να δούμε σε ποιο βαθμό αυτός ο οποίος ζητάει άσυλο καταλαβαίνει ποιες είναι οι διαδικασίες, τι αναμένεται από αυτόν ή από αυτήν και ποιος είναι ο, ο ρόλος του μέσα σε αυτή τη διαδικασία και η υποχρεώση του. Αν θέλουμε να δούμε αν είναι γνήσια μια αιτήσια ασύλου, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε σαφές προς τον ετούντα τι αναμένουμε ή τι δεν αναμένουμε από αυτόν ή από αυτήν στη διαδικασία αυτή. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με τον Προλαλήσατε ότι πρέπει να τα καταφέρουμε σωστά την πρώτη φορά. Γιατί μετά είναι πολύ πιο δύσκολο. Η μεθοδολογία για αυτές τις δύο μελέτες αφορούσε 900 ετούντες άσυλο και υπήρξε και συζήτηση σε διάφορες ομάδες. 65 <clears throat> διαφορετικές εθνικότητες καλύπτονται από την έρευνα αυτή. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι οι αιτούντες άσυλο πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τα δικαίωμά τους, δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις του, διότι υπάρχουν καταρχήν γλωσσικά φράγματα, δεν υπάρχει μετάφραση ή διερμηνία, δεν μπορούν να συζητήσουν ούτε με τους, ε, με τους δικηγόρους τους. Πολλές φορές η μετάφραση δεν λαμβάνει υπόψη τις ε, γλωσσικές τους ικανότητες. Η γλώσσα, η νομική δεν είναι κατανοητή και υπάρχει πολύ μεγάλη εστίαση στη γραπτή πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές αυτές οι πληροφορίες δεν συνοδεύονται με προφορική πληροφόρηση, ενώ η προφορική πληροφόρηση είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη αξία. Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η πληροφόρηση. Καταρχήν γιατί δίνει πρόσβαση στη διαδικασία αυτή και το άρθρο 8 της χάρτας για το δικαίωμα στην παροχή ασύλου αναφέρεται στο, στην ανάγκη πληροφόρηση. Επίσης, το Δουβλίνο 2 αναφέρεται σε περιπτώσει που πρέπει κάποιο να μεταφερθεί σε ένα άλλο κράτο μέλο, η αίτηση ασύλου. Και είναι απαραίτητο σε σχέση με τη δυνατότητα να υπάρξει προσφυγή μετά από μια άρνηση. Για την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, η πληροφορία πρέπει να δίδεται θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που δίνουν στον ετούντα τη δυνατότητα να κατανοήσει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Και αναφέρει και το θέμα των αιτήσεων βάση φύλου. Οι γυναίκες αιτούσες θα πρέπει να έχουν πληροφορία σε μια γλώσσα προσφάσιμη σε αυτήν που να τις βοηθήσει να καταλάβουν ότι μια αίτηση βάση φύλου μπορεί να είναι σημαντική σε αυτό το πλαίσιο. Για το Δουβλίνο επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν έξι χώρες ότι σε έξι χώρες αυτοί που εμπίπτουν στη διαδικασία του Δουβλίνου 2 έχουν δυσκολία σε πρόσβαση σε πληροφορία. Και δεν ξέρουν πότε θα μεταφερθούν σε κάποια άλλη χώρα ή τι θα συμβεί με την αίτησή τους. Για τις περιπτώσεις απόρριψης μιας αίτησης οι ετούντες φυσιολογικά γνωρίζουν την απόφαση αυτή, δεν ξέρουν όμως τους λόγους για την απόρριψη. Το πώς ε, γίνεται η έφεση δεν έγινε και κατανοητό. Να δούμε λίγο τη νομική κατάσταση. Τι άδες απαιτήσει γλωσσών υπάρχει πλέον στην Ευρώπη των 27. Σε 12 κράτη-μέλη. Be... Οι πληροφορίες για τη διαδικασία ασύλου θα πρέπει να διατίθεται σε γλώσσα κατανοητή για τον ετών άσυλο. Εδώ είναι τα ε, πιο σκούρα σημεία που έχετε στο χάρτη. Ε, στις χώρες που έχετε με ρίγες, ε, προσφάτως υποτίθεται ότι ε, καθορίστηκε ένα σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι τους διαθέτει γλώσσα που κατανοούν. Σε τρεις χώρες δεν υπάρχουν ε, ρυθμίσεις για τις απαιτήσεις γλωσσών βάσει νομοθεσίας. Αν δείτε τις γραπτές πληροφορίες ε, από την πλευρά του ετούντος άσυλο, σε πάνω από τα μισά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ετούντες λαμβάνουν πληροφορίες ε, είτε στη μητρική τους γλώσσα, είτε σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή για αυτούς. Σε κάποια κράτη-μέλη, λαμβάνουν πληροφορίες σε γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους, ε, κατά πάσα πιθανότητα με βάση την υπόθεση ότι θα την κατανοήσουν. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ε, μεταξύ αυτών των χωρών Υπάρχουν τρία κράτη-μέλη ε, που έχουν εθνική νομοθεσία που προβλέπει να παρέχεται πληροφορίες σε γλώσσα την οποία κατανοεί ο ετών άσυλο. Σε δύο οι ετούντε είπαν ότι λάμβαναν πληροφορίες μόνο στη γλώσσα της ε, χώρας. Αν δείτε τον αριθμό των γλωσσών ε, στις οποίες διατίθεται φυλάδια, τα οποία φυλάδια είναι ο βασικός τρόπος πληροφόρησης ε, των ετούντων άσυλο, η Γερμανία έχει τα πρωτεία με 59 γλώσσες, τη ακολουθεί η Αυστρία με 40, η Τσεχία 37 και στην άλλη πλευρά του χάρτη, στις λιγότερες ε, γλώσσες, έχουμε τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και τη Λιτωνία. Και συνεχίζουν φυσικά οι χώρες. Υπάρχουν και κάποιες χώρες ε, στις οποίες υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια νομική διάταξη που να προβλέπει μετάφραση σε διάφορες γλώσσες όπως για παράδειγμα η Δανία ε, ή το Βέλγιο που δεν έχει τόσο καλά αποτελέσματα όμως. Ο αριθμός των γλωσσών ε, θα πρέπει να συγκριθεί με τις αιτήσει ε, που κατατέθησαν το 2009 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 142 εθνικότητες το 2009. Όπως σας είπα ήδη, οι προφορικές πληροφορίες θεωρούνται πολύ χρήσιμες, ιδιαίτερα εάν ε, πρόκειται να δοθούν για να συμπληρώσουν τις γραπτές πληροφορίες που διατίθεται. Αν υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης, ε, το επίπεδο κατανόησης φυσικά είναι πολύ αυξημένο. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι ότι η ποιότητα της διερμηνίας είναι ζωτική σημασία. Now we came to the, end of the... Φτάνουμε τώρα στο τέλος της διαδικασίας, την απόφαση. Η γραπτή μετάφραση της απόφασης ε, για την παροχή ασύλου διατίθεται γραπτή ή μερική μετάφραση της γραπτής απόφασης και δεν υπάρχει γραπτή μετάφραση, αλλά πλήρης προφορική διερμηνία στις χώρες οι οποίες είναι ε, στο χάρτη ε, με ρίγες. Τα γκρίζα τμήματα του χάρτη δεν έχουν καθόλου γραπτή μετάφραση. most asylum οι περισσότεροι λοιπόν του σε άσυλο έχουν δικαίωμα έφεση ε, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά δεν έχουν πάντα πληροφορίες για νομική συνδρομή και πώς ε, μπορούν να καταθέσουν έφεση. Οι πηγές πληροφορών είναι πολύ σημαντικές και ποικίλουν ε, οι μορφές ε, παροχής πληροφοριών. Στα ε, σκούρα τμήματα της αίτησης είναι χώρες οι οποίες έχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις ως πολύ χρήσιμη πηγή πληροφόρησης. Ενώ στα κρίζα τμήματα είναι πολύ χρήσιμα τα κοινωνικά δίκτυα και έχουμε και τις λοιπές χώρες εκεί δεν μπορούσε να δοθεί καμία χρήσιμη πηγή πληροφόρησης ή δεν υπήρχε συστηματική χρήση πληροφοριών. Στις, γκρίζες χώρες, στις χώρες με ε, ρίγες έχουμε πληροφορίες από τις δημόσιες αρχές. Συμπερασματικά να σας πω ότι η γνωμοδότηση της FRA για το θέμα αυτό είναι ότι για να είναι σημαντικές ε, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται ε, τόσο προφορικός όσο και γραπτό σε μια γλώσσα που κατανοεί τον άσυλο και αυτό θα πρέπει να είναι βασική πρακτική και να θεωρείται ευρωπαϊκό πρότυπο και αυτό θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε να ε, υποστηρίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πληροφορίες τώρα για το πώς μπορεί κάποιο να καταθέσει έφεση, θα πρέπει να παρέχονται γραπτός, σε γλώσσα κατανοητή από τον ετώντα άσυλο και ή δυνατόν να του δίνονται και προφορικό οι πληροφορίες. Οι γραπτές πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε συστηματική βάση σε γυναίκες, ιδίως όταν συνοδεύονται και από άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Γυναίκες οι οποίες συνοδεύονται από το σύζυγό τους θα πρέπει να ενημερώνονται ότι μπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή αίτηση και θα πρέπει να ενημερώνονται για το δικαίωμα ε, να ε, τους γίνει συνέντευξη από άτομο του ιδίου φίλου, εάν το επιθυμούν. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις απόψεις που ήθελα να σας αναφέρω και τις αιτήσει όσον αφορά τη διάσταση του φίλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη που σας υποχρέωσα να τελειώσετε. Ξέρω ότι είναι, είναι αγχωτικό για όλους μας που πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Χωρίς αργοπορία θα δώσω το λόγο στον κύριο Κρίς Πόλετ, ο οποίος ε, θα αναφερθεί ε, σε την νομική αρρωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Δεν έχω κανέ, καμία τρομερή παρουσίαση powerpoints. θα σας τα πω έτσι με λίγα λόγια. Εγώ θα ξεκινήσω κάνοντας λίγο, ε, δημόσι, λίγο δημόσιες σχέσεις. Ε, η ΕΚΡΕ λοιπόν είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και Εξόριστων και αποτελεί την ε, συνένωση 69 μελών μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με το θέμα αυτό και δουλεύουμε για το θέμα των προσφύγων και των εξορίστων στα πλαίσια της, Ευρω... της Ευρώπης. Ε, ζητώ συγγνώμη, ε, ε, συγγνώμη, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτό το πάνελ για την έγκυρη αντιμετώπιση που είναι ένα θέμα το οποίο εδώ και καιρό μας απασχολεί και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητούμε κυρίως εδώ στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οργάνων. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εξηγήσω την άποψη του Έκρη για το front loading. Δεύτερον, θα προσπαθήσω να πω δύο λόγια σχετικά ε, με αυτό που εμείς θεωρούμε θεμελιώδες εργαλείο έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτή η έγκαιρη ε, αντιμετώπιση, αυτό το front loading στο θέμα των προσφύγων και τρίτον θα προσπαθήσω να κάνω δύο γενικές σκέψεις όσον αφορά τις προτάσεις αναδιατύπωσης της Επιτροπής. Ο Μικέλ πάρα πολύ καλά εξήγησε τι σημαίνει front-loading, έγκαιρη ε, αντιμετώπιση. Εμείς θεωρούμε ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι ε, η ε, σωστή παροχή χρημάτων, πόρων και πραγματογνωμοσύνη στο θέμα των εξορίστων και των προσφύγων και θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές από αυτούς οι οποίοι είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις και οι οποίοι έχουν τους απαραίτητους πόρους σε ό,τι αφορά την ανάγκη υποστήριξης για να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Κατά τη δική μας άποψη λοιπόν, η έγκαιρη αντιμετώπιση δεν έχει να κάνει με την ε, επιτάχυνση των διαδικασιών, γιατί όσες φορέ υπάρχει μια παρεξήγηση το θέμα αυτό. Είναι για τη βελτίωση τη ποιότητα. Και η ποιότητα μπορεί να χρειαστεί χρόνο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Συγχρόνως όμως, αν εφαρμοστεί σωστά η έγκαιρη αντιμετώπιση, αν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια μείωση του συνολικού μήκους και του κόστους της διαδικασίας παροχής ασύλου. Γιατί, γιατί οι σωστές αποφάσεις σε πρωτοβάθμιο επίπεδο μπορούν να αποτρέψουν και περαιτέρω ενστάσεις και προσφυγές. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρξουν περαιτέρω προσφυγές, αλλά αν λειτουργεί καλά το σύστημα αυτό, τότε μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες οι απαραίτητες πτυχές και αυτό θα δημιουργήσει την απαραίτητη ποιότητα. Αν ληφθεί παραδείγματος χάρη υπόψη η πληροφορία για τη χώρα προέλευση, τότε αυτό θα μειώσει το χρόνο που χρειάζονται οι δικαστέ που αντιμετωπίζουν μια μεταγενέστερη προσφυγή. Αν ο στόχο λοιπόν τη έγκαιρη αντιμετώπιση είναι να βελτιωθεί η λήψη απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Και αυτό ίσω είναι σαν να τα ξαναλέω αυτά που είπε ο Μικέλε, αλλά πιστεύουμε ότι πράγματι υπάρχουν σημαντικά στοιχεία για την ε, σωστή ε, αντιμετώπιση και αυτό βασίζεται και στην κατάρτιση αυτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά και ο φορέας του ΙΑΣΟ θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Και επίσης χρειάζεται και η παροχή νομικής βοήθειας σε αυτούς που δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν ένα δικηγόρο, γιατί αυτό είναι και επίσης και ένα στοιχείο της έγκαιρης αντιμετώπισης. Για μας σημαίνει επίσης ότι και εδώ έρχεται ένα παράδοξο όταν μιλάμε για το τέλος της, ε, για τη μείωση του μήκους της διαδικασίας αυτής, σημαίνει αυτό ότι στην αρχή της διαδικασίας χρησιμοποιείται ο απαραίτητος χρόνος για να προετοιμαστούμε για την πρώτη συνέντευξη. Για πάρα πολύ χρόνο λοιπόν έχουμε συνιστήσει στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να σέβονται τη λεγόμενη περίοδο προετοιμασίας και ανάπαυσης πριν προχωρήσει αυτή η διαδικασία, γιατί αυτό δίνει στους απαραίτητους αυτούς που ζητούν άσυλο να συζητήσουν με τον δικηγόρο τους, να συγκεντρώσουν τεκμήρια κτλ. Αυτό είναι προς το συμφέρον αυτού που ζητεί άσυλο και αλλά και προς το όφελος των αρχών οι οποίες παρέχουν το άσυλο γιατί δεν θα χάσουν χρόνο για να μπορέσουν να εξηγήσουν και πάλι στην αρχή της συνέντευξης τι πρέπει να κάνει αυτός ο οποίος έτσι άσυλο. Και επίσης μπορούν οι, οι αρχές να, να βρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη χώρα προέλευσης και να δουν αν υπάρχουν στοιχεία που κάνουν πιο ευάλωτο αυτόν που ζητάει τα, την, το άσυλο. Όλα αυτά δεν είναι θεωρητικά. Αυτή η περίοδος ε, ανάπαυλας είναι κάτι που εφαρμόζεται ήδη από, από την Ολλανδική κυβέρνηση και αυτό τώρα πια είναι τμήμα του νομικού πλαισίου στην Ολλανδία, στις κάτω χώρες. Και το Ολλανδικό Υπουργείο έχει στείλει μια επιστολή προς το Κοινοβούλιο, όπου υπάρχει αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων αυτού του συστήματος και είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να επικρίνει κανείς. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο αφορά όλους τους εμπλεκόμενους, είτε είναι ΜΚΟ, είτε είναι ε, δικηγόροι, είτε είναι ζητούντες άσυλο, ότι αυτός ο χρόνος ανάπαυλας είναι κάτι το θετικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν συζητάμε τα θέματα αυτά. Περνάω τώρα στο θέμα της ε, πρόσβασης σε δωρεάν νομική βοήθεια. Νομίζω ότι ένα σημείο κίνηση είναι το να κατανοήσουμε ότι οι διαδικασίε ασύλου στην Ευρώπη έχουν γίνει πολύ πολύπλοκε αυτός ο οποίος ζητεί άσυλο βρίσκεται σε μία μειονεκτική θέση. Γιατί δεν γνωρίζει την νομοθεσία της χώρας υποδοχής. Δεν μιλά τη γλώσσα τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό χρειάζεται βοήθεια και πιστεύουμε ότι χρειάζεται βοήθεια από την αρχή της διαδικασίας. Πιστεύουμε ότι η παρουσία στην πρώτη συνέντευξη επίσης νομικής βοήθειας είναι σημαντική είτε είναι νομομαθής, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι ε, νομικοί εμπειρογνώμονες ΜΚΟ μπορούν να βοηθήσουν να υπάρχει μια καλύτερη ποιότητα στην ε, πρώτη συνέντευξη και στην πρώτη απόφαση που λαμβάνεται για το άσυλο. Μπορούν να βοηθήσουν λοιπόν να εντοπίσουν τα ουσιαστικά θέματα και να συλλέξουν πληροφορίες, αλλά όπως βλέπουμε και στην πράξη παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών και του ετούντος. Και είναι σημαντική η εμπιστοσύνη γιατί ελλείψη εμπιστοσύνης τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι το σχέδιο για την έγκαιρη νομική βοήθεια και έχει σαν στόχο να εμπλέξει σε διαδραστικό επίπεδο τους δικηγόρους ήδη από την αρχή της διαδικασίας για την ποιότητα της διαδικασίας αυτής. Και φάνηκε και από ένα προηγούμενο σχέδιο ότι μπορούν να προκύψουν θετικά αποτελέσματα. Επειδή τελειώνει ο χρόνος, εγώ θα σας έδινα μια γενική επισκόπηση για τα πιο σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ετούντες ασύλου για τη νομική βοήθεια. Αλλά θα σας παραπέμψω σε κάποιες μελέτες. Μία από αυτές είναι μία μελέτη που κάναμε εμείς οι ίδιοι. Μία μελέτη για τη νομική αρρωγή σε σχέση με το άσυλο στην Ευρώπη, όπου κάναμε έρευνα σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 17 από τις οποίες είναι κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το θέμα αυτό της έγκαιρης αντιμετώπισης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά να πράξουμε. Αν λάβετε υπόψη το γεγονός ότι η δωρεάν νομική βοήθεια δίνεται μονάχα σε στάδιο προσφυγής σε 12 κράτη-μέλη, ενώ στα άλλα 15 υπάρχει κάποια μορφή νομικής βοήθειας στο πρώτο επίπεδο, αλλά με επικύλοντες βαθμούς και με πολλά πρακτικά προβλήματα. Όχι. Στην, στην νομοθεσία ναι, μπορεί να υπάρχει, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συστήματα τα οποία λειτουργούν και τα οποία δεν οδηγούν σε ιδιαίτερα μακροσκελείς διαδικασίες. Αυτό είναι το παράδειγμα της ε, Ολλανδίας, αλλά και στο Βέλγιο υπάρχει αυτή η προστασία και η βοήθεια. Τα κύρια προβλήματα λοιπόν που βλέπουμε είναι για την παροχή βοήθειας όταν χρειάζεται να ακολουθηθεί μια ειδική διαδικασία σε κράτη, σε επιταχυμένες διαδικασίες. Η ταχύτητα λοιπόν με την οποία γίνονται αυτές οι διαδικασίες είναι αυτή η οποία καθορίζει και δημιουργεί προβλήματα σε όλα αυτά. Για να έρθουμε σε επαφή με ένα δικηγόρο και να μπορεί κάποιο να καλέσει δικηγόρο πριν ε, επιστρέψει. Αυτό βέβαια αποτελεί πρόκληση. Για να περάσω τώρα στην τελευταία μου παρατήρηση, πάρα πολύ γρήγορα, το όλο θέμα του front-loading ε, στο πακέτο του ασύλου. Δεν ε, κρύβουμε το γεγονός ότι μας απογοήτευσαν λίγο οι προτάσεις οι οποίες κατατέθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια σειρά από θέματα τα οποία δεν είναι και τόσο φιλόδοξη για την ενίσχυση, για παράδειγμα, των προτύπων προστασίας ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το είχε αναγνωρίσει ως τεράστιο πρόβλημα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναγνωρίζουμε όμως ότι παρουσιάζονται μια σειρά πολύ σημαντικά εργαλεία για την ε, προαγωγή της προστασίας. Δεν θα τα επαναλάβω εδώ. Είναι η εκπαίδευση, είναι η προστασία στα σύνορα, η ε, ηχογράφηση των εξενεντεύξεων, ιατρικά ζητήματα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτό επίσης που διαπιστώνουμε κάνουμε είναι ότι υπάρχουν μια σειρά από διατάξει οι οποίε έχουν συμπεριληφθεί στην τροποποιημένη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υπονομεύουν αυτό το θέμα τη έγκαιρη αντιμετώπιση. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά εξυπηρετεί την επιθυμία των κρατών μελών να έχουν μεγαλύτερη ευηλιξία. Αναφέρομαι εδώ για παράδειγμα στη δυνατότητα που παρέχεται στο άρθρο 14 να υπάρχει μη εξειδικευμένο προσωπικό από άλλες υπηρεσίες ε, στην υπηρεσία ασύλου για να διεξάγει τις συνεντεύξεις. Αυτό θεωρούμε ότι είναι λανθασμένη πρακτική και αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό μακροπρόθεσμα. Ή επίσης υπάρχει η άποψη στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να μπορεί κάποιος να αναβάλει ή να μην ολοκληρώνει μια διαδικασία όταν η κατάσταση στη χώρα καταγωγής ε, του ετούντος άσολο είναι αβέβαιη και επειδή το άσυλο είναι μια προσωρινή διαδικασία, δεν θεωρούμε ότι είναι καλή πρακτική αυτή και δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη ε, να ασκούν τέτοιε πρακτικέ. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα που έχουν και να πορέχουν βοήθεια στου ανθρώπου αυτού. Ολοκληρώνοντα τώρα, επιτρέψτε μου, υπάρχει μια πτυχή που αναφέρεται στη συγκεκριμένη πρώτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την νομική αρρωγή που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα προβληματική. Είναι το θέμα ε, που αναφέρεται στο άρθρο 21, το οποίο προβλέπει αυτή τη στιγμή ότι οι νομικές διαδικαστικές πληροφορίες που μπορούν να δοθούν σε ετούντες άσυλο, καθώς επίσης και νομική αρρωγή και εκπροσώπηση στη διαδικασία της έφεσης μπορεί να δίνονται από κυβερνητικούς ε, υπαλλήλου ε, σε κρατικές υπηρεσίες. Αυτό είναι πολύ αμφισβητήσιμο κατά την άποψή μας. Θα δημιουργήσει ε, πρόβλημα σύγκρουσης ε, συμφερόντων και δεν θα έπρεπε να ενθαρρύνεται και να χρησιμοποιείται σε όλα τα συστήματα αίτησης ασύλου. Ευχαριστώ. Mm.